Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ημέρα αυτή τη μαραθώνιας Επιτροπής Αναφορών που έχουμε σήμερα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε καλά, γιατί τώρα έχουμε να ψηφίσουμε. Είναι περίπλοκη η ψηφοφορία από ό,τι μου λένε. Ελπίζω και βασίζομαι σε εσά να μην την κάνετε ακόμα πιο περίπλοκη από την απομόνη τη. Λοιπόν, ετοιμάστε τις κάρτες σε βάλτε στο μηχάνημα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Προηγουμένως όμως, πριν ψηφίσουμε, θέλω να σας ενημερώσω για τα συμπεράσματα της συνάντησης των συντονιστών που είχαμε χτες το απόγευμα. Αποφασίσαμε τα εξή. Την ημερήσια διάταξη για την Δευτέρα Ιουνίου 2016. Οι ομάδες ε, τώρα μέχρι τα τέλη του μηνός μπορούν να δώσουν στη γραμματεία άλλες προτάσεις για αναφορές όσον αφορά την ενέργεια, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Ιουλίου. Δεύτερον, όσον αφορά τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις. Το EFTD αποφάσισε να συντάξει την γνωμοδότηση όσον αφορά την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της ΕΝΒΗ για την πρόσβαση στα φάρμακα. Και η ομάδα ECR θα ετοιμάσει την γνωμοδότηση για την ΑΦΚΟ και τη όσον αφορά τη δικιά τους έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για την καλύτερη νομοθέτηση. Ευχαριστούμε. Τώρα, ό,τι στάσεις υπάρχουν ε, για τις ε, συστάσεις εγκρίθηκαν με τέσσερις εξαιρέσεις Έπειτα συζητήσαμε την ερευνη, τις ερευνητικές επισκέψεις για το 2016 και λήφθησαν δύο αποφάσεις. Πρώτον, επίσκεψη ιστορική στην Σλοβακία. 19 με 23 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη φορά που πάει στην Σλοβακία η Επιτροπή μας. Εκεί θα εξετάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναπηρία στη χώρα αυτή παρόλο που τέτοια ζητήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Αλλά είναι καλό που πάμε σε μια χώρα που δεν έχει ξαναπάει η Επιτροπή μας. Και δεύτερον θα έχουμε και ερευνητική επίσκεψη στο Ταράντο της Ιταλίας. Οκτώβριο-Νοέμβριο, την πράσινη εβδομάδα που είναι τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον στο Τάραντας. Επιπλέον, εξετάσαμε προτάσεις για μελέτες, αποφασίσαμε να ζητήσουμε μελέτες για το Linde στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης είχαμε και θέματα από τον κατάλογο Β. Οι συντονιστές σημείωσαν ότι ζήτησαν τον Μάρτιο ώστε από την B list, το B δηλαδή, να μεταφερθούν διάφορες ε, αναφορές κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα, ε, συζητήθηκαν επίσης οι κανόνες για τους ευρωβουλευτές που είναι και αναφέροντες. Συζητήσαμε με τη νομική υπηρεσία και καταλήξαμε ότι κάθε ευρωβουλευτής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως οποιοδήποτε αναφέρον. Αλλά ότι σύσταση είναι να μην συμμετέχουν στην συζήτηση για τη δικιά τους αναφορά ούτε να ψηφίζουν για τη δική τους αναφορά οι ευρωβουλευτές. Και έχουμε και την απόφαση για το 0127 του 2015. Όλοι οι ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν. Λοιπόν, δεν υπήρξε τίποτα να συζητήσουμε για το σημείο 10 που είναι τα διάφορα. Αυτά όσον αφορά την συνεδρίαση των συντονιστών και τις αποφάσεις που πήραμε εκεί. Και περνάμε στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι όσοι είναι να ψηφίσουν είναι εδώ και έχουν βάλει και τις κάρτες τους στο μηχάνημα. Ωραία, η πρώτη ψηφοφορία είναι έκθεση γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφοράς για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθεσιών. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο τίτλο από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε ποια είναι. Έχετε έτσι καλλιώ τον κατάλογο ψηφοφοριών μπροστά σα. Τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Πρέπει να διευκρινιστεί το αποτέλεσμα, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Κατά τμήματα. Το δεύτερο τμήμα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 άλλα η Πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Συμβιβαστική τρία πρώτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 4, τροπολογία 9 τώρα, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Τρίτο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 27 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Για την τροπολογία 27. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Από το ΕΛΚ ψηφίζει ένας παραπάνω από όσους πρέπει. Τώρα δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Α, εντάξει. Πέρασε τις φοφορία Εγκρίθηκε. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Το, από το ψηφίζουν ένας παραπάνω. Τώρα είναι εντάξει εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Μαριά. Και ευχαριστούμε για το έργο σας. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ο εισηγητής μας είναι η Ρόζα Στάρας Φαραγκούτ. Ψηφίζουμε λοιπόν στην συμβαστική 1 υπέρ, κατά,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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Με προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε για τη 41. Ωραία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της Εγκρίθηκε. Να το δείχνετε, να σηκώνετε τα χέρια σας, δηλαδή αλλιώς δεν μπορώ να το δω. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε και τις 47. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 48 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μήπως την 57 μέχρι την 70 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ, όχι. Α, όχι. Ωραία, μία-μία τότε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 19 τώρα. Έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από τους σοσιαλιστές για την αρχική παράγραφο της νομοδότησης. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η τροπολογία 75 καταπίπτει. Οπότε τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, την ε, Ρώσα Εστέρας. Ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε και περνάμε στη γνωμοδότηση τώρα για την 31η έκθεση όσον αφορά την παρακολούθηση και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Είναι η δικιά μου έκθεση αυτή και ελπίζω να είναι αποτελεσματική η ψηφοφορία μας. Λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Τροπολογία 6, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, θα το ελέγξουμε. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της γνωμοδότησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, περνάμε στην διερευνητική επίσκεψη στο Λονδίνο και τις συστάσεις μας. Στο Νοέμβριο ήμασταν εκεί που μας πέρασε. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Πέρας ε, της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε με διαφορά μεγάλη. Μεγάλη διαφορά. Εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, εγώ τι θέλετε να κάνω. Λοιπόν, προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και υπάρχει κατά τμήματα ψηφοφορία εδώ. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 4 με προφορική τροποποίηση. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική. Έτσι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και στη συνέχεια ψηφίζουμε το υπόλοιπο. Α, όχι. Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 5. Το υπόλοιπο καταπίπτει. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11. Με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι, ήθελα να πω εγκρίνεται λέει η πρόεδρος, άρχισα να κουράζομαι. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Συμβαστική αριθμός 1. Χωρίς την 19 τροπολογία, γιατί δεν καλύπτεται τελικά από αυτή τη συμβαστική αριθμός 1. Θα την ψηφίσουμε αργότερα. Συμβαστική 1 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 με προφορική τροποποίηση. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και το υπόλοιπο καταπίπτει. Τροπολογία 21 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Α, είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το δεύτερο τμήμα της 27. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 28. Με την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Πάλι με προφορική τροποποίηση. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στη συνέχεια, το πρώτο τμήμα, γιατί είναι κατά τμήματα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας Απορρίφθηκε. Τώρα, η προφορική 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 30. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, να ελέγξουμε και εδώ. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Τροπολογία 30, πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τέταρτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα. Αριθμός 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά πάντα, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίες εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στην διερευνητική αυτή επίσκεψη και συνεισφέρατε στην εκπόνηση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όλους όσοι θέλουν να... δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην ε, συνεδρίαση να φύγουν ήσυχα, ήσυχα από την αίθουσα και όσοι είναι να μείνουν ας ε, μείνουν για να ξεκινήσουμε με όλο το σεβασμό στους αναφέροντες που είναι παρόντες. Let's now move to, to... Μάλιστα. Ας περάσουμε στην ε, σημερινή ημερήσια διάταξη. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω το Ρούμπι Χάρολτ Κλάσον από τη Σουηδία, εξ ονόματος Σκανδιναβικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με την έκθεση για την επιμέλεια παιδιών στη Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία. Νομίζω πως η αναφέρουσα είναι εδώ παρούσα και έτοιμη να πάρει το λόγο. So, η διαδικασία λοιπόν είναι η εξή. Ε, δίνω το λόγο στην ε, αναφέρουσα για πέντε λεπτά και μετά στην Επιτροπή και στη συνέχεια στα αμέλη. Ε, δεν γνωρίζαμε ότι θα ήταν παρούσα ή αναφέρουσα, γι' αυτό πρέπει κάπως να περιορίσουμε αυτά, αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε πολλά πολλά θέματα στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Πέντε λεπτά έχετε λοιπόν στη διάθεσή σας. Chairman, πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής ε, των Αναφορών, σας χαιρετίζουμε και εξ ονόματος της ε, Σκανδιναβικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ε, μαζί με τους συνυπογράφοντες της αναφοράς 2434 του 2014, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να σας απευθύνουμε το λόγο. Πιστεύουμε ότι είναι εφαρμόσιμο το ψήφισμα ε, για την υποχρεωτική φροντίδα των παιδιών. Στείλαμε και ένα υπόμνημα στις 4 Απριλίου ε, στην Επιτροπή σας που το επιβεβαιώνει. Μετά υπάρχει ε, η υπόθεση C C435 του 2006 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ορίζει ότι ο κώδικας ε, ο ευρωπαϊκός ε, είναι εφαρμοστέος. Και η Σουηδική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως αυτή η απόφαση είναι εφαρμοστέα. Η υποχρεωτική ε, επιμέλεια των παιδιών κατά της βούλησης των γονιών και των παιδιών είναι συχνή στις σκανδιναβικές χώρες. Στη πέμπτη έκθεση της το ιε δείχνει ότι 17.000 παιδιά ε, ε, ε, τοποθετήθηκαν υποχρεωτικά σε ιδρύματα ή σε θετές οικογένειες. Ο Υπουργό ΔΕ ε, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για 20.000 παιδιά το 2014 τα οποία τοποθετήθηκαν σε ιδρύματα ή σε ανάδοχες οικογένειες. Ε, να πρόκειται για μεγάλη αύξηση ποσοστία μέσα σε πέντε χρόνια. Επενδύονται πολλά χρήματα για τις ε, ανάδοχες οικογένειες και για τα ιδρύματα. Το κόστος αυτό είναι τεράστιο και τώρα βλέπουμε μια βιομηχανία να έχει δημιουργηθεί. Απομακρύνονται τα παιδιά από τους γονείς τους και τοποθετούνται σε, θετά, σε σπίτια, σε ανάδοχες οικογένειες με αντάλλαγμα χρήματα. Ε, πρόκειται για ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά ή για απλή επιχείρηση. Βλέπουμε ποια είναι τα περιθώρια διεθνούς των διεθνών και πολυεθνικών ε, ε, εταιριών που ε, δρούν στην αγορά για την παροχή φροντίδας των παιδιών. Στη Σουηδία ε, είναι υποχρεωτική η έρευνα για τους συγγενείς ε, των ε, παιδιών. Στη Σουηδία έχει χαθεί η αίσθηση της οικογένειας, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Οι κοινωνικοί λειτουργοί προτιμούν να τοποθετούν τα παιδιά σε ανάδοχες ξένες οικογένειες παρά στους συγγενείς τους. Η κοινωνική λειτουργία και οι θετοί γονείς ε, εμποδίζουν τις επαφές ανάμεσα στα παιδιά και την πραγματική τους οικογένεια και του πραγματικούς του συγγενεί. πολλές φορές και για περιόδους 10 ετών. Είναι διαλυμένη η οικογενειακή ζωή και τα διοικητικά δικαστήρια ε, ε, επικροτούν αυτές τις αποφάσεις. Οι θετοί γονείς και η κοινωνική λειτουργή συχνά αρνούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις που είναι ευνοϊκές για τους γονείς, τους ε, πραγματικούς γονείς. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, δηλώνει ότι το κράτος θα πρέπει ε, επί να εργάζεται προς την επανένωση των οικογενειών με τα παιδιά τους και πρέπει να προσπαθούν να κρατούν τις οικογένειες μαζί και όχι να τιμωρούνται οι δικηγόροι οι οποίοι υποστηρίζουν την επανένωση των οικογενειών ή ε, μάλιστα σε κάποιες περιστάσεις η κοινωνική περιπτωσεις η κοινωνικη λειτουργια μπορει να αφαιρέσουν, να, να απομακρύνουν το δικηγόρο από την, κάποια υπόθεση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η Ντόνι Χασέν ήταν σε σε θετή οικογένεια. Η Φελίσια ε, πέθανε το 2005. Καμιά έρευνα, καμιά ανάκριση δεν έγινε. Νέα υπόθεση, η οικογένεια Μποντάρη στη Νορβηγία είναι ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται προστασία. Παιδιά και γονείς ε, αυτοκτόνησαν στις αρχές του 2015 γιατί τους αρνήθηκαν την επαφή με τους πραγματικούς τους γονείς. Θα μπορούσα να συνεχίσω με ένα σωρό περιπτώσεις. Θέλουμε να γίνει μια αποστολή Θέλουμε να δούμε αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, και δίνω το λόγο άμεσα στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, Χριστίνα Φαντιμπόκαρτ. Καλημέρα σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διεθνεί υποχρεώσει των σκανδιναβικών χωρών όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών παρακολουθούνται από του συναδέλφου μα στον ΟΗΕ. Αν δείτε το, το διαδικτυακό χώρο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, θα διαπιστώσετε ότι η Σουηδία τελευταία έχει περιοδικά εξεταστεί και όλε οι εκθέσει βρίσκονται στο διαδίκτυο της επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και ο κατάλογος σε σχέση με τη Σουηδία έχει δημοσιευθεί τελευταία. Βλέπετε την εκδοχή της 68ης Συνόδου, δηλαδή του Ιανουαρίου 2015, που δίνεται από τον ΟΗΕ, πρόκειται για αντίδραση στην κρατική έκθεση της Σουηδίας και η διαδικασία είναι εξή. Ο ΟΗΕ δημοσιεύει ένα κατάλογο ανοιχτών κρεμών θεμάτων, που θεωρεί δηλαδή προβληματικά, και ζητά από τη Σουηδία να πάρει θέση. Τώρα εγώ διάλεξα τη Σουηδία γιατί οι άλλε αναφορέ σχετίζονται στην, με τη Σουηδία, αλλά βεβαίω οι πληροφορίε αυτέ υπάρχουν για τη Φιλανδία, τη Δανία, την Νορβηγία, γιατί είναι και εκείνοι συνυπογράφουσε χώρε τη σύμβαση για το παιδί, τα δικαιώματα του παιδιού. Τι μα λέει λοιπόν ο ΙΕ για το, το Σουηδικό Σύστημα προστασία του Παιδιού και ποιε είναι τα στοιχεία που έχει για τη Σουηδία. Παραθέτω από την παράγραφο 8 του, εισέκθεση του ΑΙΕ που είπαμε βρίσκεται στον ε, διαδικτυακό χώρο. Η ΟΗΕ ζητά πληροφορίε όσον αφορά το σύστημα προστασία του παιδιού από το κράτο, ώστε να προληφθεί η ενδοοικογενειακή βία και να προληφθούν περιπτώσει κατάχρηση και παραμέληση. Ε, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι όλες οι υποθέσεις αναφέρονται εγκαίρως και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος μηχανισμός και που να είναι γνωστό στα παιδιά. Παρακαλούμε να μας δώσετε πληροφορίες κατά πόσο τα δικαιώματα ε, κατά, ε, έχουν ε, οδηγήσει σε ευξημένες διώξεις, προσφυγές από πλευρά των γονέων και αν έχει αυξηθεί η δυνατότητα των επαγγελματικών ομάδων που εργάζονται για τα παιδιά να εντοπίζουν τα παιδιά που πέφτουν θύματα βίας. Αυτά είναι τα δικαιώματα σύμφωνα με τον ΟΗΕ και όπως είπαμε ζητά από τη Σουηδία περαιτέρω πληροφορίες, επιπλέον πληροφορίες για το πώς η προλαμβάνεται η ενδοικογενειακή βία και πώς προλαμβάνεται η κατάσταση κατάχρησης και παραμέλησης παιδιών και πώς αυτή αναφέρεται. Διαβάστε επίσης τι δεν λέει η έκθεση. Η έκθεση δεν αναφέρει ισχυρισμούς και τώρα παραθέτω από τη σύνοψη της αναφοράς δεν αναφέρει ότι τα δικαστήρια δεν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους δεν αναφέρει ότι τα παιδιά υποχρεωτικά απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με καταχρηστικό τρόπο και δεν αναφέρει ότι δεν εφαρμόζεται Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ότι δεν προστατεύεται οι εγγύησεις για την οικογενειακή ζωή μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι αν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στη Σουηδία με αυτά τα θέματα, μάλλον θα είχαμε βρει κάποια αναφορά για αυτά όλα στην έκθεση του ΟΙΕ. Αλλά όχι. Και έπειτα διαρωτώμουν τι λέει ο πανεπιστημιακός κόσμος για τη λειτουργία του συστήματος επιμέλειας και πρόνοιας των παιδιών στις σκανδιναβικές χώρες και βρήκα μια ενδιαφέρουσα εισήγηση ενός καθηγητή Τάρια Πέζε του σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Τάμπερ στην Φιλανδία. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο παρουσιάζει πώς λειτουργεί το σύστημα φροντίδας των παιδιών, πρόνοιας για τα παιδιά, ενώπιον της ε, λόγου νομικών της Ιρλανδίας. Και διαβάζω εδώ ότι η πρώτη, η πρώτη ε, κοινωνική πρόνοια για τα παιδιά ε, δημιουργήθηκε στην Νορβηγία. Μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι οι σκανδιναβικές χώρε ήταν πρωτοπόρες όσον αφορά την προστασία του παιδιού. Πολύ ενδιαφέρον. Και μετά διαρωτήθηκα Επίσης, πώς ε, αντιλαμβάνονται οι μη ευρωπαϊκές χώρες ε, το πώς λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας παιδιών στις σκανδιναβικές χώρες. Ε, έκανα λοιπόν, πήγα στο, στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Προστασίας των Οικογενειών και είχαν εκεί στο site τους καλύτερη πρακτική και σχετικό παράδειγμα τη Σουηδική, το Σουηδικό Σύστημα Πρόνοιας των Παιδιών. Αναφέρονται στην Καναδά, στη Σουηδία και στο Βέλγιο και λένε ότι αν θέλετε να διαβάσουμε περισσότερα για το σύστημα προστασίας των παιδιού στην Σουηδία, βλέπουμε στο διαδίκτυο, στον χώρο της ε, αρμόδιας ε, Αυστραλιανής Επιτροπής ότι οι σκανδιναβικές χώρες έχουν έχουν ένα σύστημα πρόληψης. Αντίθετα με αυτό που έχουμε κοινό στις ε, αγγλόφωνες χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο προσανατολίζεται στην προστασία του παιδιού. Τώρα, επίσημη απάντηση της Κομισιόν. Θα ήθελα να εξηγήσω και πάλι ότι όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας για τα παιδιά στην Ένωση, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ρυθμίζεται από την Εθνική Νομοθεσία και όχι από Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 3 δεν θα επεκτείνει το, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που πρόκειται απλά για δικαιοδοσία και για επιβολή των αποφάσεων. Είναι εκτός λοιπόν του πεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πώς λειτουργούν και οι υπηρεσίε κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα για την προστασία των παιδιών. Έχουμε στοχευμένη χρηματοδότηση υπό το πρόγραμμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένειας. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα και ε, διασφαλίζουμε την αναφορά των διεθνών προδιαγραφών σε αυτά αναφερόμαστε στα αυτές τις προδιαγραφές όπως προωθούνται από τα ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και για τις, ε, τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόνοια για τα παιδιά. Όπως γνωρίζετε, για τα δικαιώματα του παιδιού έχουμε εστιάσει στο συντονισμό και τη συνεργασία όσον αφορά τα ολοκληρωμένα προγράμματα, συστήματα μάλλον προστασία των παιδιών και έχουμε προτείνει 10 αρχές για τα συστήματα αυτά που τοποθετούν το παιδί στο κέντρο και επίσης που στόχο έχουν τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους φορείς που ε, εμπλέκονται και εργάζονται για την πρόνοια του παιδιού. Η Κομισιόν καλωσορίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει αναφερθεί σε αυτές τις αρχές για την ένταξη των συστημάτων πρόνοιας παιδιού στην ε, έκθεση για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο ψήφισμα για, τα, για το συμφέρον του παιδιού που θα υιοθετηθεί σύντομα. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσει, φυσικά είμαι στη διάθεσή σα να σα απαντήσω. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την περιεκτικότατη σκιαγράφηση στοιχείων. Δεν έρχεται συχνά κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τέτοιες ε, πληροφορίες, στεγνές πληροφορίες. Όμως καλό μας κάνει πρωί-πρωί. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφου, Μάργαρετ. Αρχίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Χαίρομαι που η χώρα μου θεωρείται υπόδειγμα σε αυτόν τον τομέα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι απόλυτα αληθές. Υπάρχει μάλιστα μία ταινία αυτή τη στιγμή στη Δανία που ε, αναφέρεται στις ε, άθλιες συνθήκες επιμέλειας ε, παιδιών και τώρα οι αρχές της Δανίας ε, οφείλουν να ζητήσουν επίσημα συγγνώμη στις οικογένειε και τα παιδιά τα οποία κακοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 70 μέχρι τώρα. Ακόμα πολλές φορές στη Δανία για περιπτώσεις παιδιών που απομακρύνθηκαν και πήγαν σε ανάδοχες οικογένειε όπου μεγάλωσαν σε άσχημε συνθήκες. Εγώ ξέρω πολλά παραδείγματα και καλά και άσχημα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Σουηδία και τη Φιλανδία, όμως η Δανία δεν έχει μεταφέρει στην ομοθεσία της τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα. Ε, βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει λάθος σε όλα διότι όπως ξέρετε οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και η απόφαση επίσης δύσκολη. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να ακούσεις και τις δύο πλευρές που πολλές φορές έχουν τελείως διαφορετικά πράγματα να πούν. Και χρειάζεται φυσικά, όπως γνωρίζετε, μεγάλη προσοχή στο να αποφασίσεις ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, διότι είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένες περιπτώσεις και οι δύο πλευρές πολλές φορές έχουν δίκιο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι όλα είναι τέλεια και υπέροχα στις χώρες μας. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν νομίζω πως έχουμε βρει μία λύση στο θέμα αυτό δεν νομίζω πως η αυστηρή νομοθεσία που έχουμε είναι απόλυτα σωστή, όπου οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν προτεραιότητα στην ανατροφή ενός παιδιού, στη Δανία τουλάχιστον. Υπάρχουν, όπως σας είπα, πολλά παραδείγματα που έχουν γίνει λάθη και είναι δύσκολο να πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο δεν μπορώ να καταλάβω ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση εάν η αρμοδιότητα είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στη χώρα μου, όμως έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί τα γεγονότα δεν μπορώ να το δεχτώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Κύριε Μαρτάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω ακριβώς τη θέση να κρατήσω. Ακούω και την Επιτροπή, ακούω και τους αναφέροντες που θέτουν κάποια ζητήματα. Νομίζω ότι αυτά που θέτουν φαίνονται να μην ισχύουν. Ακούω όμως τι λέει και η Επιτροπή. Συνήθως οι περιπτώσεις που φτάνουν σε εμά είναι τραγικές. Ψηφίσαμε μία έκθεση σχετικά με τη μελέτη που κάναμε τον Νοέμβριο, την έρευνά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ακούω ότι θα πάμε και στη Σλοβακία, όπου να είναι. Και μετά, ποιος θα έχει σειρά. Γιατί ακούμε για τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των γονιών, που τελικά υπάρχουν σε όλες λίγο πολύ τις χώρες. Οπότε μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μία έρευνα συνολικά για το ζήτημα αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω φυσικά το δίκαιο στη Δανία, στη Σουηδία, πώς ακριβώς έχει. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι προσέχουμε, ακούμε τους αναφέροντες, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να αναλύσουμε το θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλό θα ήταν να μας πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Για να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή τη θητεία. Σα ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ρομπέρτο. Ευχαριστώ. Ακούω τους συναδέλφους που λένε ότι είναι πολύ λεπτές υποθέσεις. Και αφορούν πάρα πολλές οικογένειες. Και όχι μόνο οικογένειες, αλλά και τον περίνα της κοινωνίας μας. Άκουσα την ε, αναφορά, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο θα ήθελα να σταθώ στο ότι χρειάζεται μια ανάλυση των ε, διεθνών τυχών αυτής της αναφοράς. Αναφέρομαι στις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής και στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. κοιτάζοντας το Βρυξέλλες 2α, τίνω να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δηλαδή αναφέρεται σε θέματα δικαιοδοσίας και επιβολής αποφάσεων. Αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Δεν είμαι πεπισμένη για το αν οι αναφορές αυτές είναι αρκετά σχετικές έτσι ώστε εμείς να πρέπει να αναλύσουμε το αν έχει γίνει παράβαση του κανονισμού ή όχι και να δούμε επίσης αν ο κανονισμός εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση. Χρειάζεται επίσης να δούμε εάν και κατά πόσο μπορεί να ε, αφορά και την περίπτωση της Νορβηγίας. Ο συνάδελφος κύριος Μαρτάν πρότεινε να κάνουμε μια διερευνητική αποστολή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα κράτη-μέλη και να κοιτάξουμε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι χρειάζεται να συζητηθεί το θέμα και να δούμε πώς τα δικαιώματα ε, του παιδιού θα ε, συνδυαστούν με τις δικές μας αρμοδιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιτέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την κυρία Μετσόλια. Πέραν αυτού όμως, η αναφέρουσα δεν απέδειξε ότι το θέμα έχει σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ε, περίπτωση της ε, Δανίας, η οποία διαπραγματεύτηκε και κέρδισε ένα opt-out. Ούτε μπορεί να εφαρμοστεί στην Νορβηγία, διότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βρυξέλλες 2α μπορεί να εφαρμοστεί στην Σουηδία ή τη Φινλανδία, όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση αφορά επιβολή δικαστικών, ε, εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Και τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν για τις προϋποθέσεις και τους ε, όρους που διέπουν την απομάκρυνση ενός παιδιού και την τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια. Η δική μου λοιπόν πρόταση είναι να κλείσει αυτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπαν πολλοί συνάδελφοι ήδη και ε, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό θέλω να, σας, ε, να το μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς, ε, αυτή η Επιτροπή των Αναφορών λαμβάνει όλο ένα, ε, πάντοτε μάλλον μεγάλο αριθμό αναφορών που αφορούν την ευημερία των παιδιών. Και αυτό είναι λόγος μεγάλης ανησυχίας. Καλούμεθα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις πώς θα μπορέσουμε να παρέμβουμε. Όμως η κατάσταση η ίδια, αυτή καθ' αυτή, ε, προσωπικά είναι πολύ λυπηρή και δραματική. Κάτι που με εντυπωσίασε στην ε, παρουσίαση της αναφέρουσας ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, ε, δηλαδή μίλησε για business. Αυτό πραγματικά μου φαίνεται πολύ ανησυχητικό και Αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η πραγματικότητα τη στιγμή που έχουμε τόσο διαφορετικές ε, απόψεις και πόσο δύσκολο είναι για αυτή την Επιτροπή να προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως δίνει τη δική της εκδοχή, κάνει την εργασία της. Ε, βλέπουμε, ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες να, βρεθούν, ε, να βρεθεί κοινό τόπος. Τη στιγμή που οι εθνικές νομοθεσίες είναι τόσο διαφορετικές και μάλιστα πολλές φορές είναι δυσνόητες για μας που εδώ προσπαθούμε να δώσουμε μια όσο γίνεται πιο ομοιόμορφη ε, εικόνα. Εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι στο να προσπαθήσω να προχωρήσω με αυτές τις αναφορές. Ε, δικιά μας ε, καθήκον σε αυτή την ομάδα εργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θα κοιτάξουμε εκ νέου να εξετάσουμε αυτές τις ε, υποθέσεις. Ε, Αντί λοιπόν να γίνει μια μελέτη που μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο, καλύτερα ίσως θα είναι να διοργανώσουμε μια εκδήλωση με συμμετοχή των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων ε, των κρατών μελών. Ε, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, μια πρόταση που θα ήθελα να κάνω για την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, για την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και μαζί για να κατανοήσουμε πώς θα μπορέσουμε προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Thank you, Eleonora. Ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο προ το παρόν, γι' αυτό θα δώσω ξανά το λόγο στην αναφέρουσα. Έχετε δύο λεπτά. Ονομάζομαι Elizabeth Σέιφερ και συνεργάζομαι με την ε, κυρία Κλάξον στην Επιτροπή αυτή. Ως ε, δικηγόρος εργάζομαι πέντε χρόνια. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι από το 1930 στη Σουηδία έχουμε υπηρεσίες παιδικής μέρημνας από το κράτος. Έχουμε κάπως τροτσκιστικό τρόπο θεώρησης της οικογένειας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θεωρούνται μέρος της οικογένειας αλλά μέρος της κοινωνίας. Επομένως τα δικαιώματα των παιδιών δεν είναι συνδεδεμένα με την οικογένεια και με το σπίτι. Τα δικαιώματα των παιδιών αφορούν την κοινωνία και το κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα παιδικής ε, μερίμνας από το 1930. Στη Σουηδία η οικογένεια για μας δεν συνδέεται με θρησκευτικές πεπιθήσεις. Συνήθως σε περιπτώσεις απομάκρυνσης παιδιών ε, πηγαίνουν δύο αστυνομικοί και δύο κοινωνικοί λειτουργοί στο σπίτι που θα, από το οποίο θα απομακρυνθεί το παιδί. Και μάλιστα σε μία περίπτωση είχαν έρθει, είχε έρθει η αστυνομία με χειροβομβίδες κρότου και η γυναίκα από την οποία απομάκρυναν το παιδί ήταν μια μητέρα παιδιού πέντε μηνών. Τη πήραν όμως το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη Σουηδία. Έρχονται πολλές φορές και μας ζητούν βοήθεια νέες μητέρες και πολλές φορές η κατάληξη είναι να χάσουν το παιδί τους. Τα χρήματα δηλαδή δεν ε, εξοδεύονται για το καλό του παιδιού και πολλές φορές μάλιστα απομακρύνουν τα παιδιά από ε, μητέρες που τα μεγαλώνουν μόνες τους. Και αυτή η τάση είναι πολύ έντονη στη χώρα μας. Τώρα μάλιστα έχουμε πολλές περιπτώσεις απομάκρυνσης παιδιών από μετανάστες αυτές οι οικογένειες χάνουν τα πάντα όταν χάσουν το παιδί τους. Χάνουν οποιαδήποτε ε, κοινωνική παροχή, χάνουν επιδόματα στεγαστικά κτλ. Και μιλάμε για ποσά ύψους 40.000 ε, κορονών το μήνα για κάθε παιδί. Είναι λοιπόν μεγάλο το πρόβλημα και πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα θέμα που αφορά καθαρά ε, τις ε, χώρες ε, αυτές και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α αναφέρεται σε θέματα δικαιοδοσίας και εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και δεν υπάρχει κάποια διασυνοριακή πτυχή που να ρυθμίζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Δανία, όπως ακούσαμε, είναι εξαίρεση, αποτελεί εξαίρεση γιατί έχει επιλέξει opt-out. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν ο κανονισμός αυτός αφορά τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα, διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε ως Επιτροπή Αναφορών είναι να παραπέμψουμε το θέμα στην ομάδα εργασίας για την παιδική ημέρημνα, την οποία προεδρεύει η κυρία Εύη, το οποίο θα μπορούσαν να το εξετάσουν και να το εξετάσουν με έναν τρόπο δημιουργικό, να δουν ποια νέα στοιχεία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προτού λάβει χώρα η αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Προτείνω λοιπόν να ευχαριστήσουμε καταρχάς τους ε, αναφέροντες που ήρθαν και μας παρουσίασαν την αναφορά και να παραπέμψουμε το θέμα στην ομάδα εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Μπορείτε να δεχτείτε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε από τη Σουηδία στις Βρυξέλλες. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Αναφορά 2453 Ολλανδία σχετικά με την απομάκρυνση των παιδιών από την Νάνση Σχάουτεν. Η αναφέρουσα δεν βρίσκεται σήμερα εδώ. Δεν ήρθε. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως ε, από ό,τι μου είπαν η αναφορά δεν ε, εστάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Τότε θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους αν επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Εντάξει, αν χρειαστεί θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια γιατί έχω διαβάσει την αναφορά, λέει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Διάβασα λοιπόν την αστυνομική έκθεση η οποία αναφέρει ότι τα παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα στο δωμάτιό τους με μεγάλη ποσότητα ούρων και δυσοσμίας εκεί. Αναφέρεται επίσης ότι το δικαστήριο της Σουηδίας δεν ήταν αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση διότι τα ε, παιδιά δεν ε, είχαν σουηδική υπηκότητα. Ωστόσο δεν μας έχει σταλεί αναφορά αυτή και δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν ε, καταφέρα να διερευνήσω την υπόθεση. Όπως σας είπα δεν λάβαμε κάποια πληροφορία σχετικά με την αναφορά. Επομένως δεν μπορώ να κρίνω την ε, αρμοδιότητα ή όχι που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν όντω το Σουηδικό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, τότε αλλάζει το θέμα. Θα έπρεπε όμως να δω την απόφαση του δικαστηρίου προτού σχολιάσω οτιδήποτε παραπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως μας είπατε δεν έχετε λάβει τον φάκελο της υπόθεσης. Ωστόσο γιατί, εφόσον δεν έχετε λάβει τίποτα, έχουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η εξήγηση θα μπορούσε να είναι απλή. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ζήτησε να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κάτι το οποίο θεωρώ ανόητο, μια και δεν έχουμε τον πλήρη φάκελο να αποστείλουμε στην Επιτροπή. Η αναφέρουσα δεν βρίσκεται εδώ. Δεν έχουμε έγγραφα τα οποία να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους για να μου προτείνετε πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Η κυρία Πιτέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε την πλήρη τεκμηρίωση για να εξετάσουμε το θέμα. Η έκθεση αυτή της αστυνομίας είναι φοβερή τώρα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες για τις εκθέσεις αστυνομίας, πάντως αυτά είναι τα γεγονότα όπως τα αναφέρει η αστυνομία και δεν είχε επιλογή, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει τίποτα άλλο. Ας περιμένουμε λοιπόν τα υπόλοιπα έγγραφα πριν προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το εξή. Πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή γιατί η έκθεση της αστυνομίας είναι τόσο τρομερή. Έχουμε τόσες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την μέρημνα των παιδιών. Εγώ εκτιμώ προκαταρτικά ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει το να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Τι λέτε εσείς συνάδελφοι, συμφωνείτε να την κλείσουμε. Ναι, ναι. Ναι. Α, κυρία Όκεν. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ακόμα και την Ορβηγία την αφορά, Μάργαρετ. Νομίζω ότι εσείς είστε στην προηγούμενη αναφορά. Έχουμε περάσει στην επόμενη. Εγώ λέω για την επόμενη αναφορά. Οι συνάδελφοι εδώ με στηρίζουν να κλείσουμε την αναφορά. Βλέπω ότι το ΕΛΚ, το FD, το ECR να γνέφουν καταφατικά και οι σοσιαλιστές. Οπότε κλείνουμε αυτή την αναφορά και περάμε στην επόμενη αναφορά που είναι η αναφορά 1140 του Hans Jespersen, δανικής ηθαγένεια σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, πάλι στη Δανία και τη Σουηδία. Δεν είναι εδώ αναφέρον. Όπως και έγινε και με την προηγούμενη περίπτωση, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι στην ημερήσια διάταξη, γιατί ένας συνάδελφος από την Επιτροπή μας ζήτησε να μπει στην ημερήσια διάταξη. Λυπούμε λοιπόν που το λέω, αλλά είναι στην εμμυρίσια διάταξη, είναι πολύ γενική, ό,τι αναφέρεται εδώ είναι κάτι πολύ γενικό, δεν πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επιπλέον πληροφορίες ότι υπάρχει εδώ μάλλον σύγχυση δημιουργεί. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ορθολογικά αυτή την αναφορά. Εφόσον όμως ένα συναδερφός ζήτησε να μπει στην εμερήσια διάταξη, δίνω το λόγο στους συναδέρφους. Και σας ζητώ να με συμβουλέψετε πώς να συνεχίσουμε με την ε, αναφορά αυτή. Ρομπέρτα, τι λες. Δεν ξέρω πόσο μπορώ να βοηθήσω, αλλά συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που έχουμε στη θέση μας είναι πολύ περιορισμένες. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να την κλείσουμε ή να την αφήσουμε ακόμα ανοιχτή μέχρι να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν ξέρω τι διαδικασία, δηλαδή τι παραπάνω πληροφορίες χρειαζόμαστε για να τις συζητήσουμε. Αν δεν τις πάρουμε να την κλείσουμε τότε. Αλλά μας κάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως αποφασίσουμε όντας ε, εν γνώση των γεγονότων και όχι έτσι. Μαρλένα. Συμφωνώ. Πρέπει να την κλείσουμε γιατί δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Ε, μάλλον νομίζω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και μετά να την κλείσουμε. Ελονόρα, Κι εγώ. Συμφωνώ. Ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Θα μπορούσαμε να πάμε το θέμα στην ομάδα εργασίας για τα δικαιώματα του παιδιού, να έχουμε την εκτίμηση κάποιου εμπειρογνώμονα. Συμφωνώ, λέει η πρόεδρος, ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ να προτείνω, να την αφήσουμε ανοιχτή, να την στείλουμε στην ειδική ομάδα και όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δούμε. Συνεχίζουμε με την αναφορά 0171. Ε, Γερμανική ηθαγένεια είναι μια αναφέρουσα εξ ονόματος της Animals Angels με πάρα πολλές υπογραφές σχετικά με τη μεταφορά ζών των ζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ η αναφέρουσα. Η Κρίστα Μπλανκέ λοιπόν έχει το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, πριν από δύο εβδομάδες ένα γερμανικό φορτηγό από τον Λίβανο ήρθε με διάφορες, ε, διάφορα βοηδή. Ήταν υπερφορτωμένο, δεν ήταν καλά κλειστή πόρτα, δεν υπήρχε αρκετό νερό και υπήρχαν ε, δύο μικρές αγελάδες που ε, γέννησαν μοσχαράκια. Το ένα πέθανε. Πριν από δέκα μέρες πήρε φωτιά κάπου στην Ιταλία και πέθαναν δέκα ζώα. Τέτοια γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά στην Ευρώπη. Η ρύθμιση 1205 δεν μπορεί να εμποδίσει τέτοιου είδους ε, γεγονότα. Η σύσταση της Επιτροπής πάντα είναι ότι αν εφαρμόζονται καλύτερα οι κανόνες όλα θα είναι μια χαρά. Τα πράγματα όμως δεν ε, αλλάζουν επειδή κάποιος επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια για 10 χρόνια. Εγώ σας έχω δώσει τα σχετικά έγγραφα στις ε, 204 σελίδες του κειμένου μας αποδεικνύουμε ότι έτσι όπως έχει σήμερα η ρύθμιση είναι αδύνατο να προστατεύονται τα ζώντα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Το έγγραφο αυτό απορρέει από 20 χρόνια εμπειρίας στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Είναι ότι καλύτερο έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή για την μεταφορά των ζώντων ζώων. Δεν θα επαναλάβω τα στοιχεία που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να σας μιλήσω για τους ανθρώπους, παρόλο που εγώ είμαι ακτιβίστα για την προστασία των ζώων. Οι αστυνομικοί είναι εκείνοι τελικά που πρέπει να θέτουν σε εφαρμογή μια ρύθμιση η οποία είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Για 20 χρόνια λοιπόν η Animals Angels, η οργάνωσή μας, έχει συνεργαστεί με την αστυνομία έχει σταματήσει φορτηγά, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σωρό καταστάσεις στους δρόμους. Μερικές φορές τρεις η ώρα το πρωί μας σε ένα αστυνομικό τμήμα για να δούμε τι έχει γίνει σε έναν ισπανικό αυτοκινητόδρομο. Η αστυνομία μας έχει ζητήσει και έχουμε βοηθήσει με επιμόρφωση τους αστυνομικούς, έχοντας οργανώσει διάφορα εργαστήρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά τους και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άδικη όταν τις δικές της τις ευθύνες για την εγγύηση της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά τους την βάζει στους ώμους των αστυνομικών οι οποίοι δεν έχουν καν τα μέσα για να εφαρμόσουν την νομοθεσία, τη ρύθμιση ούτε για τον χρόνο μεταφοράς, ούτε μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. Οπότε σκεφτείτε τους αστυνομικούς κάθε φορά που μιλάτε για επιβολή του νόμου. Η επιβολή του νόμου δεν είναι κάτι αόριστο, έχει να κάνει με ανθρώπους και με τους περιορισμούς που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τα δύνατα δυνατά από τους αστυνομικούς και σίγουρα όχι τώρα που έχουν και άλλα θέματα όπως είναι τρομοκρατία και μετανάστευση. Για να μην υποφέρουν τα ζώα λοιπόν και για να μην υπερφορτώνονται οι αστυνομικοί, θα σας ζητούσα να αφήσετε ανοιχτή την αναφορά αυτή και να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι καλύτερο από το να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να τηρεί τον νόμος. Το 1991 η Επιτροπή Αναφορών πήρε μια μυστορική απόφαση όταν εξέτασε αναφορά με χιλιάδες υπογραφές που ζητούσε την αναγνώριση της ευημερία των ζώων. Οι συνάδελφοί σας τότε ε, φρόντισαν να υπάρξει και αλλαγή στη συνθήκη. Και σήμερα μπορείτε κι εσείς να κάνετε ένα εξίσου μεγάλο βήμα υπέρ της ευημερία των ζώων όταν αυτά μεταφέρονται. Την αναφορά μου την στηρίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογράφοντες και από τους περισσότερους ευρωβουλευτές, οι κτηνίατροι στην Ευρώπη και στις χώρες ε, μέλη Δανία, Γερμανία ζητούν έναν περιορισμό στο χρόνο μεταφοράς των ζώων των Κάτι πρέπει να σημαίνει δημοκρατία. Οπότε σας εκλυπαρώ, κρατήστε την αναφορά αυτή ανοιχτή. Το θέμα της μεταφοράς ζώων των ζώων έχει τεράστια σημασία για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και η μόνη μας ελπίδα είσαστε εσείς κυρία Πρόεδρε και τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, για την παρουσία σας εδώ και για τις ανησυχίες σας που μας εκφράσατε. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, τον κύριο Ντένι Σιμονίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να πω το εξή. Να επαναλάβω καταρχήν δυστυχώς όσα επαναλαμβάνουμε και εμείς στην απάντησή μας που είναι παλιά. Λοιπόν, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για νέα νομοθεσία γιατί πιστεύει ότι είναι ένα ζήτημα σωστής εφαρμογής του νόμου. Αυτό που μπορώ συμπληρωματικά να πω, γιατί από το 2012 ε, διάφορα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπενθυμίζω ότι η εφαρμογή του νόμου είναι θέμα αρμοδιότητας των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να δουλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, να ενσωματώνουν τον νόμο δηλαδή. Και στα πλαίσια αυτά, από το 2011 που είχαμε έκθεση για τη μεταφορά των ζώων, ξεκινήσαμε διάφορες δράσεις. Υπήρξαν παρεμβάσεις στις χώρες μέλη για τον ρόλο τους στην Ειδική Επιτροπή που έχει να κάνει με τη μεταφορά των ζώων και την διατροφή τους. Δύο φορές το χρόνο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει συνάντηση με τα εθνικά σημεία επαφής που είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες στις χώρες μέλη που ασχολούνται με ειδικά θέματα εφαρμογής του κανονισμού, κάτι το οποίο έχει δώσει πολλά αποτελέσματα μέχρι τώρα στις χώρες μέλη υπήρξε και τροποποίηση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της για να βελτιώσει τις εκθέσεις που γίνονται μετά από ελέγχους. Επίσης, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα ειδικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό του 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πειραματικό αυτό πρόγραμμα που ισχύει για τρία χρόνια με σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μεταφοράς των ζώων. Συμφωνώ απόλυτα με την αναφέρουσα για το ότι το θέμα της εφαρμογής είναι θέμα που έχει να κάνει με ανθρώπους. Άνθρωποι εφαρμόζουν τον νόμο, πράγματι. Και δεν είναι με την υιοθέτηση νόμων που έχει να κάνει για παράδειγμα με το χρόνο μεταφορά στο ζώων λύνονται όλα. Μακάρι, αλλά δεν ισχύει αυτό δυστυχώς. Το θέμα του χρόνου μεταφοράς δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε, όπως είπε και η αναφέρουσα, είναι θέμα και συνθήκων μεταφοράς θερμοκρασίες κλπ. Οπότε μαζί όντω πρέπει να φροντίζουμε για την επιμόρφωση των ανθρώπων που δουλεύουν επί τόπου. Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο, αλλά γι' αυτό Πρέπει να υπάρχει συνοχή στη δράση μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι συνάδελφοι, ποιος θέλει το λόγο, Μαρλένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ πρέπει να πω ότι η ιδιότητά μου είναι αντιπρόεδρος στην Δικαινοβουλευτική Επιτροπή για την Ευημερία των Ζώων. Οπότε έχω ίδιο συμφέρον, ας πούμε. Αν δείτε κάτι ταινίε που δείχνουμε στις συνεδριάσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά των ζώων, πώς βασανίζονται, πώς υποφέρουν, τότε νομίζω ότι όλοι θα φροντίζαμε να διασφαλίσουμε ότι συμμόρφωση θα υπήρχε, που δεν υπάρχει τώρα. Όντως, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση. Το λειτουργικό έργο δεν φτάνει. Τα ζωντανά αυτά υποφέρουν. Οπότε δεν μας κάνουν τα επιχειρήματα τα νομικίστικα που λένε ότι είναι θέμα εφαρμογής του νόμου, συμμόρφωσης, επιβολής κτλ. Αυτά δεν μας οδηγούν πουθενά. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με ε, κουτιά ξύλων ε, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλων προϊόντων που είναι άψυχα, έχουμε να κάνουμε με έψυχα ζώα, με ζώντα ζώα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάει ακόμα πιο μακριά από το θέμα το καθαρά νομικό της νομοθεσίας δηλαδή. Ελεονόρα, επόμενο μιλήτρια. Ευχαριστώ. Και εγώ Πιστεύω ότι πρέπει να μην ανοιχτή αυτή η αναφορά για έναν απλούστατο λόγο, διότι μας θυμίζει ότι παρά το ότι στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουμε τα ζώα ως έμψυχα ε, ζώα που έχουν ε, αισθησή, ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό δεν συμβαίνει, διότι δυστυχώς ε, όπως λέγαμε και πριν τα μεταχειρίζονται ως εμπορεύματα, ως προϊόντα και αυτό το θυμόμαστε και στη φάση που αναφερόμαστε στους κανόνες ε, που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά ζών των ζώων, θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι την τελευταία περίοδο έχουμε δραματική αύξηση των ορών ε, ταξιδιού των ζώων και κυρίως αυτό το οποίο σε έλεγε και πριν η Κομισιόν, υπάρχει και αυτό η συλλογή στοιχείων και ελπίζω πως θα είναι αποτελεσματική, αλλά μέχρι στιγμής σίγουρα είναι ελληματική. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε να ξανά προτείνουμε εντόνως τη θέσπιση ενός ε, ορίου ταξιδιού, ε, ορών ταξιδιού, 8 ε, ορών. Αυτή τη στιγμή τέτοιο όριο δεν υπάρχει και αυτό είναι εις βάρος των ζώων. Πιστεύω πως σίγουρα το θέμα των ελέγχων και της παρακολούθησης που γίνεται από πλευράς των κρατών μελών και των επιθεωρητών, δηλαδή ολόκληρη η υπόθεση των ανθρωπίνων πόρων που χρησιμοποιούνται προφανώς θα πρέπει να εμβαθυνθεί. Ε, πιθανότατα θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, αναφορά ανοιχτή και να τη στείλουμε και στο περιβάλλον, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ώστε να κάνουν και εκείνη μια γνωμοδότηση και να προτείνουν και πάλι ένα όριο όριο ε, ορών μεταφοράς των ζωντανών ζώων. Ευχαριστώ. Πίτερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτείνω να ακολουθήσουμε την πρόταση να συμπεριλάβουμε και τις αρμόδιες επιτροπές. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και έχουμε συζητήσει το θέμα και εκεί. Ε, πιστεύω όμως ότι στην Επιτροπή Γεωργίας τουλάχιστον δεν είχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν έχω πρόβλημα ε, επίσης ε, με τον ε, ορισμό ζώα εκτροφής. Σίγουρα όμως πρέπει να φροντίζουμε η μεταφορά να είναι σωστή, η μεταφορά των ζώων και στα σφαγεία. Τώρα, σχετικά με το χρονικό περιορισμό. Πιστεύω πως πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Η πρόταση για ανώτατο όριο 8 ωρών ε, για μένα είναι σωστή. Θα μπορούσαμε μάλιστα να μειώσουμε ε, το όριο αυτό, να κάνουμε ακόμα λιγότερες ε, τις ώρες τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταφέρονται ζώα τη φορά. Και σίγουρα οι έλεγχοι θα έπρεπε να εφαρμόζονται καλύτερα. Ο χρόνος μεταφοράς λοιπόν πρέπει να οριστεί, πρέπει να περιοριστεί. Άλλο ένα πρόβλημα είναι και η έλεγχη. Εδώ πιστεύω πως πρέπει να ζητήσουμε και τη συνδρομή της Επιτροπής Μεταφορών για να κοιτάξουμε τις ανισορροπίες. Γίνονται πολλοί έλεγχοι στις εθνικές οδούς, ξέρετε, σε ε, φορτηγά αυτοκίνητα, όμως αυτή η έλεγχη ε, είναι εστιασμένη αλλού, στο ωράριο των ε, οδηγών, αλλά όχι στις συνθήκες μεταφοράς των ζώων. Πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να έχουμε όχι περισσότερους ελέγχους, καλύτερους ελέγχους, καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο όταν θα σταματά τα φορτηγά για έλεγχο να κοιτάζει όχι μόνο τι γίνεται στην καμπίνα του οδηγού αλλά και πίσω από αυτόν. Πώς ε, ταξιδεύουν τα ζώα, σε τι συνθήκες. Πώς είναι ο εξοπλισμός που τους παρέχει νερό, τροφή. Είναι λοιπόν ε, πολύ χρήσιμο να ζητήσουμε τη συνδρομή και της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Γεωργίας και όλων των επιτροπών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτή η πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ε, Ζώων Εκτροφής και η Συνθήκη της Λισαβόνας ε, καθιστούν σαφές ότι τα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλη αξία. Η προστασία των ζώων είναι κοινωνικό ε, γεγονός, κοινωνικό κανθήκον είναι κάτι που δείχνει την κοινωνία αξιών μας, δείχνει τις αξίες μας ή την έλλειψη αυτών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνεται και από το πώς συμπεριφέρεται στα ζώα. Κρίνεται και από τον πρωτοπόρο ρόλο ή όχι που αναλαμβάνει στην προστασία των ζώων. Συμμετείχα την ε, περασμένη εβδομάδα στο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία των ζώων και εκεί συζητήθηκε το θέμα της ε, μεταφοράς τους. Αυτό που συνειδητοποίησαν όλοι είναι ότι η μεταφορά των ζώων γίνεται υπό απαράδεκτες συνθήκες. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και σοβαρές ελλείψεις τους ελέγχους, περιπτώσεις ε, κακομεταχείρισης. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί το χρονικό όριο μεταφοράς των ζώων και σίγουρα η Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα καθώς και η Επιτροπή Μεταφορών. Αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στα ζώα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο αξιών, αλλά το οφείλουμε και στους ίδιους μας, ε, τους εαυτούς ως άνθρωποι, διότι τα ζώα είναι όντα ζωντανά που αισθάνονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι συγκεντρώθηκαν ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Αυτό σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι υπέγραψαν και ακόμα περισσότεροι αρνούνται αυτή ε, την ε, μεταχείριση των ζώων, αυτόν τον βανσανισμό των ζώων. Αυτό που είναι κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ε, αρνητική κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει το δικαίωμα στα ακροδεξιά κόμματα να ανθίσουν, να μεγαλώσουν με τις πράξεις μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια τελευταία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήσει τα λόγια και να προβεί επιτέλους σε πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Το, το λόγο έχει η κυρία Χάουσεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καθημερινά εκατομμύρια ζώα σφάζονται στην Ευρώπη. Χιλιάδες χιλιόμετρα διανύουν μέσα σε κακές συνθήκες για να φτάσουν στα σφαγεία. Όμως τα ζώα είναι τα ζώα τα ζώα τα οποία εξετάζουμε και που αναγνωρίζει την ευημερία τους η νομοθεσία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτά. Εδώ πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει την αναφορά αυτή. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και αλλού, όλοι αυτοί ζητούν να αλλάξει η ρύθμιση για τη μεταφορά των ζών των ζώων. Εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας. Είχαμε μια γραπτή δήλωση στο παρελθόν. Και είχαμε πει ότι το δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει όχι μόνο για τη μεταφορά μέσα στην Ευρώπη αλλά και εκτός. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λέει ότι έχει βοηθήσει σε κάτι λίγο, δεν έχει αλλάξει όμως πραγματικά τη ρύθμιση. Καθημερινά, λοιπόν, περιμένουν τα ζώα στα σύνορα με την Τουρκία για ώρες και μέρες. Μεταφέρονται, αποδυναμώνονται, είτε πρόκειται για ζώα που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα, είτε πρόκειται για νεογέννητα. Θα έλεγα λοιπόν, πηγαίνετε στα σύνορα αυτά, πηγαίνετε να δείτε τι συμβαίνει. Το είπε και η συνάδελφός στη κοινοβουλευτική ομάδα στο Στρασβούργο ότι είδαμε διάφορα φιλμάκια με αυτή την τραγική κατάσταση. Πραγματικά είναι να σπαράσει καρδιά σου άμα δεις πώς βασανίζονται αυτά τα ζώα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα. Μα τι περιμένουν. Λέω λοιπόν, η μεταφορά των ζών των ζώων, εφόσον είναι αναγκαίο να γίνεται, πρέπει να κρατάει λίγο και να υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός με κανόνες που εφαρμόζονται. Θα ήθελα λοιπόν αναθεώρηση της ρύθμισης, μια πρόταση δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να αναθεωρεί την ισχύουσα ρύθμιση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και έτσι κλείνει ο κύριος ομιλητών όσον αφορά την αναφορά αυτή και δίνω το λόγο και πάλι στην αναφέρουσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο δύσκολο για μένα να προσθέσω κάτι, γιατί είναι η πρώτη φορά, βλέπετε, που είχα την ευκαιρία να τα ακούσω όλα αυτά από εσά. Συνήθω μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μα ακούει ποτέ. Δέκα χρόνια τώρα. Και τώρα αυτά που είπατε εσεί πραγματικά έφτασαν κατευθείαν στην καρδιά μου. Τα καλά σας λόγια, η κατανόηση που δείχνετε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και για μένα είναι συγκινητικό που σας ακούω να το λέτε αυτό, γιατί ακριβώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει φορτωθεί πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να φτιάξει καταρχήν αυτήν την ε, ομάδα για την ευημερία των ζώων και οι συνάδελφοι πρέπει να ξέρετε ότι οι ίδιοι βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν και οι υπόλοιποι που δεν ασχολιόντουσαν με τέτοια ζητήματα το τι ακριβώς συμβαίνει και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και για την γενοδορία σας και για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ και για το ότι συμπάσχετε με αυτά τα όντα που υποφέρουν. Ολοκληρώνουμε λοιπόν. Φυσικά και θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και σημειώνουμε και αυτό που είπε και ο Πίτερ ότι δηλαδή πρέπει να συμμετάσχει εδώ και η Επιτροπή Μεταφορών, γιατί δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα. Συνεπώς, θα στείλουμε την αναφορά αυτή και την τεκμηρίωση που διαθέτουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή Γεωργίας. Θέλω επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε στην Επιτροπή μας με την αναφορά αυτή. Οπότε ίσως δεν σας προσκαλέσουμε ξανά Ξέρουμε, ξέρετε μάλλον εσείς ότι εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αναφορά σας. Δεν θα σας αναγκάσουμε να ξανάρθετε στις Βρυξέλλες. Μάλιστα δεν είναι και τόσο εύκολο να φτάσει κανείς στις Βρυξέλλες στις μέρες μας. Να είσαστε όμως σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Αναφορών, ασχολείται με την αναφορά σας. Αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχατε στη συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι ε, πολλές αναφορές όσον αφορά την απαγόρευση της τελετουργικής σφαγής ζώων. Πάλι έχει να κάνει με την ευημερία των ζώων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά είναι ένα πιο περίπλοκο θέμα αυτό. Θα δώσω λοιπόν... Α, ο αναφέρον δεν είναι εδώ. Το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύς αμέσως. Παρακαλώ. συγγνώμη, είχα, είχα αφοσιωθεί εδώ, είχα απορροφηθεί. Λοιπόν, στην ουσία, εδώ αναφέρω να ζητά στο κανονισμό του, για, την θανάτωση ή την σφαγή υπάρχει μια απαγόρευση της τηλετουργικής σφαγής ζώων για την με, με, με ζάλι. Ε, ε, αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι ο κανονισμός σήμερα εκφράζει ένα κάποιο επίπεδο ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των ζώων που όντως έχει γραφτεί στη συνθήκη στο άρθρο 13 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης το άρθρο 10 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης που αναφέρεται στην ανεξιθρησκεία. Μέχρι στιγμής ε, ανέκαθεν υπήρχε και αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ε, ότι υπάρχει αυτή η εξαίρεση αλλά ότι τα κράτη-μέλη ε, είναι αυτά που την εφαρμόζουν και ότι ο κανονισμός αναγνωρίζει μια κάποια ευελιξία ή πάση περιπτώσει κάποιο περιθώριο ερμηνείας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις για την τελετουργική σφαγή τη στιγμή που αυτό γίνεται σε σφαγείο. Ε, δεν έχουμε στόχο, σκοπό να αλλάξουμε αυτές τις διατάξεις γιατί πιστεύουμε ότι κατοπτρίζουν μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πτυχές της ε, συνθήκης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, οι συνάδελφοι μπορούν τώρα να πάρουν το λόγο. Η κυρία Άουκεν. That Νομίζω πως θα πρέπει να σκεφτούμε αν το ζώο υποφέρει ή όχι. Γιατί τι είδου προσευχές και ό,τι και αν κάνουν, δεν νομίζω πως το ζώο ενδιαφέρεται γι' αυτό και ούτε και εμένα θα με ενδιαφέρει να σα πω την αλήθεια. Εφόσον το ζώο υποφέρει και εδώ έχουμε προβλήματα με τα μεγάλα ζώα και το πιστόλι ζάλης, γιατί αν δεν το χρησιμοποιηθεί αυτό σωστά, στη Δανία α πούμε ξέρω και έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω τώρα πώ γίνεται, ότι οι μουσουλμάνοι δέχτηκαν στην σφαγή χαλάλ να χρησιμοποιήσουν το πιστόλι ζάλης ε, μέσα στο πλαίσιο της τελειτουργικής σφαγής για ένα μεγάλο ζώο ένα μεγάλο ζώο παίρνει πολλή ώρα να χάσει τις αισθήσεις του όταν απλά τα αφήνουν να ε, χάνει το αίμα του σιγά σιγά εφόσον κάτι απαγορεύεται σε μια χώρα δεν πρέπει να επιτρέπεται μόνο και μόνο για θρησκευτικού λόγους όχι, δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Αλλά εάν το έχουμε και στα, στη θανάτωση σφαγή πτηνών και τα λοιπά και εξάχων και τα λοιπά. Είναι, δεν έχει να κάνει τίποτα με την θρησκεία αυτό που συμβαίνει. Ο βιομηχανικός τρόπος με τον οποίο γίνεται ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω απλά να ακούσω τι, πόσα παραδείγματα έχουμε στην Ευρώπη για κράτη-μέλη που επιτρέπουν τη σφαγή μεγάλων ζώων χωρίς κανένας είδους ε, ζάλι. Στην αργή δηλαδή ε, ε, την απώλεια του αίματος χωρίς κανένας είδους αναισθησία. Πίτερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για μένα είναι ντεζαβού αυτό, διότι το 2003 ήδη ασχολήθηκα στο Εθνικό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό και ήμουν ειδικό ε, απευθεμελός της ομάδας μου γι' αυτό. Παρατήρησα πόσο γρήγορα κάποιος περνά από τα μικρά θέματα στα μεγάλα όταν ασχολείται με αυτά. Εμείς στην αρχή, ξέρετε, είχαμε μια ξεκάθαρη ε, γραμμή. Λέγαμε ότι το ζώο πρέπει να έχει αναισθητοποιηθεί πριν τη σφαγή. Αυτό ήταν κοινή παραδοχή. Και μετά όταν μπήκαμε στη, στα, μεγάλα, στα βαθιά νερά της πολιτικής, τότε άρχισαν και εμφανίζονταν διάφορες διατάξεις, διάφορες παρεκκλήσεις και άρχισε να συζητιέται και το θέμα της ε, ζάλης. Ίσως ε, έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα στους ε, θρησκευτικούς κύκλους. Υπάρχουν ορισμένοι κύκλοι που βλέπουν το θέμα με κάποιες ε, αμφιβολίες. Εδώ δεν πρόκειται, πιστεύω, να, για την απαγόρευση της ε, πρακτικής αυτής, αλλά για κάποια αναισθητοποίηση του ζώου πριν τη σφαγή. Χρειάζεται, πιστεύω, μεγάλη προσοχή και χρειάζεται να δούμε και τις ε, λεπτομέρειες. Όταν λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει και να το κάνουμε. Στις ε, στον τελετουργικό τρόπο σφαγής ε, τα ζώα πρέπει να μην έχουν τις αισθήσει τους, όπως απαγορεύεται γενικότερα. Πιστεύω πως ε, θα ήταν κρίμα να κλείσουμε αυτή την αναφορά προσωπικά διότι το θέμα δεν έχει λήξει. Σας λέω, ασχολούμαι προσωπικά εδώ και 15 χρόνια με αυτό και δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Το θέμα δεν είναι βέβαια ότι ε, πρέπει να συζητηθεί, αλλά το πώς πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και πρέπει να παραμερίσουμε τα συμφέροντα, πρέπει να δούμε την προστασία των ζώων και να σταθούμε σε αυτό μόνο, σε αυτόν τον στενό ορισμό. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος για το φόρουμ που πρέπει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χέρζενκαμ. Ευχαριστώ. Στην Ολλανδία δύο εκατομμύρια ζώα περίπου κάθε χρόνο ε, σφάζονται με αυτόν τον τρόπο. για τις εβραϊκές αγορές και τις ε, ισλαμικές αγορές. Μόνο στην Ολλανδία, έτσι. Ναι, δεν εξαίρεση. Η Ολλανδία σε όλη την Ευρώπη κάτι αντίστοιχο έχουμε. Η επιστημονική έρευνα είναι σαφής ότι εφόσον θανατώνονται χωρίς νάρκωση προηγουμένως τα ζώα, αυτό είναι κάτι το οποίο τα κάνει να υποφέρουν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν είναι απαράδεκτο για μας. Και είναι για την ελευθερία της θρησκείας, αλλά η ελευθερία αυτή πρέπει να σταματάει όταν αρχίζουν να υποφέρουν τα ζώα οι άνθρωποι. Για μένα, βάσει του συντάγματος των χωρών μελών, αλλά και της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά και της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, νομίζω ότι πρέπει να πετήσουμε να γίνεται η νάρκωση δεν είναι κάτι που ταιριάζει με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Δεν μπορεί οι θρησκείες να οδηγούν σε θύματα. Είτε πρόκειται για την, ευρωπαϊκή, για την εβραϊκή θρησκεία, είτε τη μουσουλμανική. Στην Ολλανδία είχα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες στο Εθνικό Κοινοβούλιο πριν από μερικά χρόνια. Δυστυχώς δεν προχώρησε τίποτα, κυρίως εξαιτίας της διαμαρτυρίας της εβραϊκής κοινότητας εκεί. Είναι σημαντικό, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιάρ, να γίνει η συζήτηση. Για μένα, εντάξει, δεν χρειάζεται να κλείσει, μπορεί να παραμείνει προς συζήτηση το θέμα και θεωρώ ότι είναι κρίμα που η Επιτροπή Γεωργίας απλώς στέλνει μια επιστολή αντί να καθίσει και να συζητήσει σε βάθος το θέμα. Όπως και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζώα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να πάρει κάποια πρωτοβουλία για το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να τονίσω πως ε, ότι φυσικά η, σφαγή, τελετουργική σφαγή, η σφαγή χωρίς ανασυντοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, διότι πολύ εύκολα μπορούν να σε χαρακτηρίσουν αντισημίτη ή αντιμουσουλμάνο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα να απαλλαγή από τις ε, θρησκευτικές πτυχές του. Η τελετουργική σφαγή για τα ζώα προκαλεί ε, μεγάλο πόνο. Και ακριβώς επειδή έχουμε υπογράψει τις ε, ευρωπαϊκές, τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των ζώων, είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόσουμε. Θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο. Ε, το Πανεπιστήμιο του Καΐρου αναφέρει ότι η σφαγή με αναισθητοποίηση δεν τηρεί τις ε, προδιαγραφές που ορίζει το Κοράνιο. Και η Αίγυπτος είναι μια μουσουλμανική χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πραγματικότητα η απαγόρευση της αναισθησίας κατά τη σφαγή των ζώων. Υπάρχει πολιτική θέληση γι' αυτό. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και τι γίνεται εκεί. Μήπως θα μπορούσαν κάποιες άλλες χώρες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, όπως ε, δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Τουρκία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να συζητήσουμε το θέμα άλλη μία φορά δημόσια, όμως με τον αναγκαίο σεβασμό προς τις ε, θρησκευτικές κοινότητες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ε, Πολύ σύντομα. Ε, Είμαι ευχαριστημένη από την συζήτηση έτσι όπως γίνεται τώρα και νομίζω πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε έναν κοινό τόπο. Σίγουρα τα ζώα δεν ενδιαφέρονται, όπως σας είπα, για προσευχές, για λειτουργίες κτλ. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για το εάν ακόμα στην Ευρώπη γίνεται σφαγή ζώων χωρίς αναισθησία. Διότι είμαι σίγουρη ε, ότι το σκεπτικό του ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ε, πιστόλι ζάλης έχει να κάνει με αυτήν την ε, τελετουργική σφαγή. Και σίγουρα μπορώ να καταλάβω την ε, οπτική γωνία αυτών που θυσιάζουν τελετουργικά ζώα, και εντάξει δεν μπορείς να πας να θυσιάσεις ένα μισοπεθαμένο ζώο. Όμως, αυτά που σκέφτομαι ή πρεσβεύω εγώ δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα εφαρμόσω και σε μια νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί για το καλό των ζώων, για να μην αισθάνονται πόνο και να μην υποφέρουν τα ζώα την ώρα της φαγής. Είναι κάποια κατάλοιπα από απαρχαιωμένα συστήματα, κάποια κατάλοιπα επίσης θρησκευτικά και πιστεύω ότι όταν μπλέκουμε τη θρησκεία με το καλό των ζώων τότε οδηγούμαστε λίγο σε ένα θέατρο του παραλόγου. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, άρα θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα και προτείνω το εξή. Μόλις με ενημέρωσαν ότι το τμήμα πολιτικής πολύ σύντομα, σε μερικές εβδομάδες ή το πολύ μερικούς μήνες, θα εκπονήσει μια νέα μελέτη για, την, για το ευζοία των ε, ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και μόλις παρουσιαστεί η μελέτη, εμείς ως Επιτροπή να αναλάβουμε την διοργάνωση μιας εκδήλωσης όπου θα καλέσουμε και τις άλλες αρμόδιες επιτροπές και όλους τους ενδιαφερόμενους και θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τη μελέτη μελέτη για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής σχετικά με την ευζοία των ζώων, η οποία έληξε το 2015 και το τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτό το χώρο, όμω αναγνωρίζω ότι σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει και δεν μπορούμε να ρίχνουμε το βάρο μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει και εμεί να αναλάβουμε δράση για να προχωρήσει το ζήτημα. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου πρόταση. Τη δέχεστε? Ναι. Ωραία. Έτσι θα πράξουμε λοιπόν. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω κάποιους από εσάς που μπαίνουν μέσα και μου θυμίσα την επόμενη αναφορά, δηλαδή την κοπή της ουράς των ε, χείρων στη Δανία. Έχουμε λοιπόν μία αναφορά για αυτό ακριβώς το θέμα. Μάλλον τρεις αναφορές. Και θα δώσω το λόγο στους αναφέροντες. Όλγα Κίκοφ, ε, αναφορά 721 και άλλη μία. Πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Η αναφορά είναι από το HSI Η αναφορά αυτή αναφέρεται στην ε, συνεχή κοπή της ουράς των χείρων. Η οδηγία του 2008 όμως αναφέρει διάφορα πράγματα μέσα και ένα από αυτά ε, λέει ότι οι χείροι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αρκετό υλικό, σε δραστηριότητες δηλαδή, και στην ίδια οδηγία προβλέπουμε την απαγόρευση της ε, τακτικής σκοπής των ε, ουρών των χείρων και ότι πριν φτάσει κανείς σε αυτό το μέτρο πρέπει να πάρει άλλα μέτρα για να αποφύγει τα ζώα μεταξύ τους να δαγκώνονται. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες και το 2008 και το 2009 πήγαμε στη Γερμανία, τη Δανία, την Ουγγαρία, τις κάτω χώρες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ερευνήσαμε και σε διάφορες ε, φάρμες. Το 2013 επίσης πήγαμε στην Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία. Είδαμε λοιπόν ότι πάνω από 90% των χείρων πέραγαν από αυτή τη διαδικασία κοπής των ουρών τους και ότι πάρα πολλοί χείροι δεν είχαν στη διάθεσή τους ε, το υλικό το οποίο προβλέπει η οδηγία. Και επειδή δαγκώνται μεταξύ τους οι χείροι, γι' αυτό οι κτηνοτρόφοι τους κόβουν την ουρά. Όμως, η οργάνωσή μας είπε ότι ο κυριότερος λόγος που δαγκώνουν τις ουρές τους είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή, αρκετό υλικό για να απασχολούνται. Το θέμα αυτό του εμπλουτισμού των υλικών δεν είναι το μόνο, η πρόσβαση δηλαδή σε επαρκή ποσότητα υλικών δεν είναι το μόνο. Ε, ο σανός είναι ένα από τα καλύτερα, τα ασφαλέστερα τρόφιμα και χρησιμοποιείται ε, σαν υλικό εμπλουτισμού, αλλά είδαμε ότι αυτό συμβαίνει σε πολύ λίγες εκτροφικές ε, μονάδες. Ο εμπλουτισμός ε, των, ε, της τροφής είναι επίσης κάτι που κρατάει τα ζώα απασχολημένα και είδαμε ότι σε ορισμένες μονάδες υπάρχουν και άλλα υλικά που είναι ανακατεμένα με τον σανό. Εδώ σε αυτό το πίνακα βλέπετε ότι ο σανός είναι το καλύτερο, το άχυρο είναι το καλύτερο υλικό για να αποφεύγεται το δάγκωμα ε, της ουράς και βλέπουμε ότι και άλλες μέθοδοι με κάποια αλυσίδα, με κάτι πλαστικά παιχνίδια δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά, για να μην πω δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά. Διάφορα μέτρα μειώνουν το κίνδυνο του δαγκώματος πέρα από τον εμπλουτισμό αυτών σε υλικά, η κατάλληλη τροφή, ε, να έχουν νερό, το κλιματικό περιβάλλον που είναι καλό για τα ζώα. Υπάρχει το θέμα της υγείας, το να είναι σε καλή υγεία τα ζώα, να μην ανακατεύονται πολύ μεταξύ τους και να χωρίζουμε τα θύματα από τους θύτες, τους χείρους δηλαδή που δαγκώνουν ρες από τα υπόλοιπα ζώα. Κατά το παρελθόν, από το 2003, η έχει υποβάλει διάφορες εκθέσεις όσον αφορά το φαινόμενο αυτό και το πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κοπή της ουράς. Διάφορα μέτρα έχουν ληφθεί υπόψη από τον κλάδο και τους κτηνοτρόφους. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να εφαρμοστεί η οδηγία. Το 2014, το Μάρτιο πιο συγκεκριμένα, είχαμε 470.000 ε, αναφορές που πήγανε στην ε, Επιτροπή και 59 ευρωβουλευτές ζήτησαν να εφαρμόζεται ορθά η οδηγία. Πριν από ένα μήνα η Κομισιόν εξέδωσε σύσταση για μέτρα προκειμένου να μειωθεί η κοπή της ουράς. Συγχαρητήρια λοιπόν από εμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπέβαλε τις συστάσεις αυτές. Όμως, οι κανόνες υπήρχαν για χρόνια και δεν εφαρμόζονταν. Οπότε, κτηνοτρόφοι και ο κλάδος γνώριζε τα μέτρα που μπορούσαν να πάρουν ε, για να μειωθεί το φαινόμενο. Τα μέτρα αυτά όμως δεν τα εφάρμοζαν. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε τώρα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και τα κράτη-μέλη είναι να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις αυτές και να φροντίσουν όλες οι χώρες μέλη, όλες οι πλευρές να φροντίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα. Θέλουμε επίσης να δούμε και ένα χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του νόμου. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα θέλαμε οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο. Και θέλουμε να έχουμε και τη δυνατότητα της διαδικασίας επί παραβάση, προκειμένου να δίνουμε κι εμείς κάποια συνέχεια, γιατί αλλιώ θα παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση. Δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα. Τη στιγμή που ο νόμος υπήρχε έτσι καλώς τόσα χρόνια και δεν εφαρμόζονταν, Μόνο αν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία κυρώσεων, μόνο τότε ε, υπάρχει περίπτωση για κάποια πρόοδο. Thank you. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή. Μόλις ενημερώθηκα για το ότι έχουμε τη μελέτη του τμήματος πολιτικής ΓΑΜΑ. Υπάρχει εδώ στην αίθουσα. Οπότε παρακαλώ και στους, στις αναφέρουσες παρακαλώ και σε όλους να τη δώσετε. Πολύ φρέσκια. Σας ε, προτρέπω να την μελετήσετε όλοι. Λοιπόν, τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σιμονή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, γνωρίζω τη μελέτη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοπή της ουράς των χείρων. Πολύ καλή ποιότητα, δεν το λέω αυτοπίσημα, το λέω προσωπικά. Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πραγματικά πολύ καλή. Η Επιτροπή λοιπόν συνυπογράφει απόλυτα στα όσα παρουσίασε η αναφέρουσα ότι δηλαδή υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα με τις σχετικές ρυθμίσεις και γι' αυτό και προχώρησε σε συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συμπληρώσω όμως ότι η σύσταση συνδέεται και με μια ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επίσης έχει εκδώσει κάτι με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάει για πολύ συγκεκριμένες λύσεις και εναλλακτικά. Τώρα, ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν παθιάζει το αν θα βάλουμε ψανό ή αν θα σταματήσουμε να κόβουμε τίσουρες. Γιατί τα λέμε αυτά, γιατί το πρώτο που χρειάζεται είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Η διατροφή, η πρόσβαση σε υλικά, είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα δηλαδή και απαιτεί γνώσεις και διάδοση της πληροφορίας. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που δημοσιεύτηκαν οι συστάσεις μας θα φροντίσουμε να κυκλοφορήσουν επαρκώς να γίνουν γνωστές όχι μόνο στις χώρες μέλη αλλά γενικότερα στην αγροτική κοινότητα γιατί όντως πολλές φορές δεν είναι γνωστές οι εναλλακτικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει και διάφορες δράσεις. Ήδη υπάρχουν τρεις επισκέψεις μελέτης σε τρεις που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές. Έχουμε πάρει εθνικούς εμπειρογνώμονες με τους οποίους ε, επισκεπτόμαστε την Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ελβετία που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές ακριβώς για να ενημερωθούν οι πυρογνώμονες από τις χώρες μέλη. Τρεις τέτοιες επισκέψεις λοιπόν έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς και επιπλέον αλλά αυτό γίνεται πιο συχνά. Έχουμε κάποιες ε, ενημερωτικές ε, ε, συναντήσεις για επιμόρφωση όσον αφορά την ευζοία και πιο συγκεκριμένα και για τους χείρους. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ήταν η τελευταία φορά και επικεντρωθήκαμε ακριβώς σε αυτό το θέμα, πώς δηλαδή να εφαρμόζεται η σύσταση. Αυτά είναι όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς πιστεύω ότι πράγματι θα έχει ένα πιο λεπτομερές πρόγραμμα δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε όπως ζήτησε και η αναφέρουσα να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με, γιατί όχι, δυνατότητες δράσης περισσότερο δεσμευτικές αν αυτό κρυθεί αναγκαίο, αλλά εξαρτάται από το πώς θα εκτιμηθεί η κατάσταση. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα μπορείτε να πάρετε το λόγο αν θέλετε. Η Μάργαρετ. Øh. Ναι, είναι μια πολύ δανέζικη υπόθεση, γι' αυτό θα μιλήσω δανέζικα. Ορισμένοι από εσά θα θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει όλα αυτά ε, από το 2014 ήδη Είχαμε συζητήσει, είχαμε πάει επί τόπου, είχαμε συνομιλήσει με τη Σουηδική και Δανέζικη και τηλεόραση και είχαμε μιλήσει για αυτές τις πρακτικές στις χώρες. Ε, με αυτή την υπόθεση λοιπόν πολλοί άνθρωποι παρακολούθησαν την υπόθεση από Δανέζικης και Σουηδικής πλευράς και οι καταναλωτές στην Σουηδία ακόμα και αν το κρέας ήταν πιο ακριβό μποϊκοτάρισαν το δανέζικο χοιρινό κρέας ή έκαναν συστηματικά κοπή τη ουρά των χείρων. Οι καταναλωτέ επέλεξαν δηλαδή την ευημερία των ζώων, ακόμα και αν αυτό κοστίζει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είχε άμεσα θετικό, άμεση θετική επίπτωση. Αλλά βεβαίω αυτό χρειάζεται ε, τακτικά ε, εκστρατείε και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό από πλευράς ε, της ε, Κομισιόν για να εφαρμοστεί πραγματικά η ε, κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, κάπως γνωρίζω την υπόθεση αυτή, έχουμε, την έχω μελετήσει, ποιες είναι οι συνθήκες εκτροφής στις μονάδες και μέσα στις κλοβούς Δεν γίνεται ε, όπως σε, βιομηχανικό επίπεδο να κρατώνται τα οι Και μάλιστα είναι πολύ πιο απαιτητικοί οι σε σχέση ας πούμε με τα σκυλιά. Ε, μπορεί να, ζει, να παίξουν ας πούμε με δύο-τρεις μέρες αλλά μετά το βαριέται. Υπάρχει βέβαια το άχυρο, χρειάζονται οι χείροι μια διασκεδαστική ε, ζωή Er Αν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να τρώμε χοιρινό κρέα, θα πρέπει να διερωτηθούμε πώ θα τα εκτρέφουμε τους χείρου. Στη Δανία χρησιμοποιείται πολύ το χοιρινό. Γι' αυτό και είναι προς το συμφέρον μας να ζουν καλύτερα. Ε, υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού. Πρέπει να αποφευθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Γι' αυτό και θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να ξαναδεί την έκθεση και να προχωρήσει η διαδικασία. Να γίνει μια διαδικασία κατά παράβαση εναντίον των χωρών που δεσέβονται την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Και... Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Η κοπή της ουράς των χείρων είναι μια διαδικασία που πονάει. Την ε, έχουμε αποδεχτεί για να αποφεύγεται το δάγκωμα της ουράς από άλλους χείρους. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να βρούμε τρόπο να αποφύγουμε. Το είδαμε και στην παρουσίαση. Βέβαια, όταν βρίσκονται μέσα σε ένα κακό περιβάλλον ε, οι χείροι, πάρα πολύ και δεν έχουν ε, άλλη δυνατότητα. Κάτι ακούστηκε για μεταλλικές μπάλες. Ναι, ε, γιατί σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να παίζουν οι χείροι με τέτοιες μεταλλικές μπάλες Όμως είναι αφελές αυτό. Όπως είπε και η κυρία Όκεν, είναι έξυπνα ζώα οι χείροι. Και χρειάζονται κάτι που να τους τραβά την προσοχή. Ένας πιο φυσικός τρόπος, με περισσότερο σανό, με εμπλουτισμένο υλικό, για να μπορούν να συμπεριφέρονται και αυτά φυσιολογικά όπως είναι στη φύση τους. Τώρα εδώ έχει χαρτογραφηθεί ένα πρόβλημα το οποίο ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στην Ευρώπη. Από το 2003 έχουν γίνει διάφορες έρευνες, διάφορες εκθέσεις και κάθε φορά το συμπέρασμα είναι ότι δεν φτάνουν οι σημερινοί κανόνες, ότι παραβιάζονται. Η Επιτροπή λέει, μα υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύσαμε, Ωραία, είναι ένα καλό βήμα αυτό, ένα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση για να σταματήσει αυτή η συστηματική κοπή της ουράς των χείρων. Όμως, το πραγματικό πρόβλημα έχει να κάνει με την εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η έκθεση, πολύ καλή. Όμως, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε με περισσότερη ένταση να φροντίσει να επιδιώξει τη διαδικασία επί παραβάση για κυρώσει σε βάρος όσων δεν συμμορφώνονται. Η διαφορά ποια είναι με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και την προηγούμενη ρύθμιση. Αν δεν εφαρμόζονται, Είναι λοιπόν ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάποια κρόση. Ευχαριστώ, Ελεονόρα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω να προσθέσω έναν γενικότερο προβληματισμό που αφορά τη χρήση των ε, ζώων στις εντατικές ε, ε, μονάδες και αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το ότι αυτό το μοντέλο εντατικής εκτροφή είναι απαράδεκτο. δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις διατάξεις των του άρθρου 13 για την, της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τα ζώα είναι έμψυχα ε, και το επαναλαμβάνω για τον απλό λόγο ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους στο, στην κτηνοτροφία και στη γεωργία έχει φτάσει σε φερικτά επίπεδα είναι το παράδειγμα του πιο τρελού καταναλωτισμού, γιατί πάρα πολλά από τα ζώα που εκτρέφονται τελικά καταλήγουν ως ε, διατροφικό απόβλητο και δεν τρώγονται καν. Εγώ προσωπικά δεν ε, τρώω κρέας, ε, εδώ και πολλά χρόνια προσέχω, και γι' αυτό και με απασχολούν πολύ αυτά τα θέματα και κατά κάποιο τρόπο καταγγέλλω αυτό που είναι μια γενική συμπεριφορά της κοινωνίας που είναι πολύ παράδοξη. θα έπρεπε όλα αυτά να γίνονται για να αυτό που θα έπρεπε να γίνει μάλλον για την προστασία όχι μόνο των ζώων αλλά και τη, τη, τη, δική μας υγεία των ανθρώπων ε, ήταν μια δραστική μείωση κατανάλωσης του κρέατος. Κάθε φορά Ακούμε ε, αδύναμο, ε, μάλλον θεωρούμε ότι είναι αδύναμο επιχείρημα, ενώ αντίθετα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραλαμβάνουμε κάθε φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι από αύριο πρέπει να κλείσουν όλες οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αλίμονο, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όντω να προβληματιστούμε ευρύτερα. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίω αυτό που λείπει ω συνήθω είναι η σωστή εφαρμογή των κανονισμών και ελπίζω ότι με αυτή την αναφορά που θα πρέπει να μείνει άνοιχτη για να κατά κάποιο τρόπο να διατηρήσουμε μια πίεση για τη σωστή εφαρμογή, να δώσουμε συγκεκριμένε ε, ημερομηνίε για να εφαρμοστούν οι κανόνε που πρέπει να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει και μια ομοιόμορφη αγορά. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Μαλέν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα ισχυριστώ ότι είμαι ειδικό τους χείρους και, θα, και πώς ξέρω πώς να τα σταματήσω να δαγκώνουν τις ουρέ τους. Όμως ε, καταλαβαίνω πως είναι βάναυσο το να κόβονται οι ουρές τους. Πιστεύω πως εδώ έχουμε θέμα εφαρμογής και επιβολής νομοθεσία και σίγουρα δεν είναι δύσκολο να ελέγξουμε όχι όλα τα εκτροφία, αλλά τουλάχιστον αρκετά, όσα τουλάχιστον εφαρμόζουν αυτήν την ε, πρακτική. Και το πιο εύκολο πιστεύω πως θα ήταν να συμπεριλάβουμε και τους καταναλωτές εδώ, οι οποίοι θα κληθούν να αναλογιστούν ναι, αν θα έπρεπε εκτός από το κρέας να υπάρχει και πληροφορία πάνω στο πακέτο για το αν αυτό το κρέας έχει προέλθει από εκτροφία τα οποία ε, εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές. Και θα μπορούσαμε επίσης να προωθήσουμε ε, εκείνους οι οποίοι συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Πάντως αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε κάτι τόσο Βάναυσο. Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά που είπε η Ελεονόρα Εύη. Ο κτηνοτρόφος παράγει αυτό που του ζητείται από την αγορά. Και όταν ο καταναλωτής αλλάζει τη συμπεριφορά του και ζητά άλλα προϊόντα, τότε και ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης θα προσαρμοστεί αναλόγως. Τα τελευταία δέκα χρόνια δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία βελτίωση ως προς την ευζοία των ζώων και θα μπορούσαμε ίσως ε, να ζητήσουμε πιο έντονα ε, να γίνουν βελτιώσεις. Αυτό το έχουμε δει στην περίπτωση της εκτροφής βοηδών. Έπειτα, στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό έχουμε απαγορεύσει το, την εκτροφή βοηδών δεμένα. και την μεμονωμένη εκτροφή, διότι τα βόδι είναι γελαία ζώα και πρέπει να έχουν ε, και άλλα ζώα του είδους τους μαζί. Τώρα, πιστεύω πως η νομοθεσία σε γενικές γραμμές είναι καλή. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, δεν έχουν πρόβλημα ε, οι νόμοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε έτσι με πολύ ωραία λόγια ότι η διαδικασία ε, παραβάση είναι κάτι ε, που αποτελεί καλή ιδέα, όμως το θέμα είναι ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Δεν ξέρω λοιπόν εάν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι καθόλου το πόσο χρήσιμη θα ήταν μια τέτοια διαδικασία. Αυτό που θα έλεγα είναι να φροντίσουμε τους νόμους. Εάν δεν θέλουμε την κοπή της ουράς των χείρων, τότε πρέπει να το απαγορεύσουμε. Και πρέπει να δημιουργηθούν μέτρα και προδιαγραφές για το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Στην τελική πρέπει να διαλέξουμε εάν θα ανεχτούμε αυτές τις πρακτικές ή εάν θα τις απαγορεύσουμε. Σίγουρα όπως ε, αναφέρθηκε υπάρχει και θέμα στρέβλωσης του ανταγωνισμού, διότι κάποιοι εφαρμόζουν τον κανονισμό, κάποιοι όχι, κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα προσωπικά να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή, έτσι και αλλιώς υπάρχει και μελέτη, μπορούμε και να απευθυνθούμε στην ε, αρμόδια Επιτροπή για περισσότερη βοήθεια. και θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάποιο χρονικό περιθώριο, για παράδειγμα δύο χρόνια ή δέκα χρόνια, για να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αλλά ας περιμένουμε τη μελέτη για να δούμε και περισσότερες πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς, οι εμπειρογνώμονες αυτή τη στιγμή εργάζονται έτσι ώστε να βοηθήσουν εμάς. Θα δούμε λοιπόν, να περιμένουμε τα στατιστικά στοιχεία και τη μελέτη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά γεγονός είναι ότι οι πράξεις και λόγια διαφέρουν πάρα πολύ. Μαργκρέτα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι υπάρχει νομοθεσία, αλλά δεν μπορούμε να την εφαρμόζουμε κατά το δοκούν. Οι νόμοι πρέπει να είναι σεβαστοί από όλους και να εφαρμόζονται συστηματικά. Αυτή η συστηματική κοπή της ουράς των χείρων είναι παράνομη και συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζεται εν μέρη λόγω των συνθήκων στις οποίες εκτρέφονται τα ζώα. Ε, δεν νομίζω ότι οι μικρές φάρμες είναι η καλύτερη λύση. Πιστεύω ότι και μια μεγάλη φάρμα μπορεί να παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ε, στα ζώα αυτά. Αν δείτε πώς συμπεριφέρονται τα ζώα όταν είναι έξω στη φύση, τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Οι αγελάδες, για παράδειγμα, έχουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά αν έχετε δει χείρους έξω στη φύση, ε, θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι η συμπεριφορά, ο εγκλισμός τους αυτός ε, στις, ε, στους μικρούς χώρους στα ε, εκτροφία. Το να τηρούνται οι νόμοι δεν είναι μόνο ε, κάτι το θεωρητικό. Όταν τηρούνται οι νόμοι έχουμε και καλύτερο κρέας στο πιάτο μας. Καλύτερη ποιότητα. Και όταν η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν εφαρμόζει τους νόμους, τότε αυτό ναι, αποτελεί διαστρέβλωση του ανταγωνισμού και αθέμητη πρακτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τους αναφέροντες. Έχετε δύο λεπτά. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε όλα αυτά τα σχόλια και συμφωνούμε πολύ με ναι, όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τι έχει γίνει από το 2003 μέχρι τώρα. Από το 2003 υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη μέτρων για να απαγορευτεί η κοπή της ουράς των χείρων. Και αυτά τα μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί. Η νομοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί από του αγρότες, από του κτηνοκτρόφους. Όπως σας είπα, πάνω από το 90% των εκτροφίων που είδαμε και κοιτάξαμε εκατοντάδες εκτροφία, ε, έκοβαν τις ουρές των χείρων. Είναι λοιπόν κάτι που είναι μια εγχείρηση ρουτίνας για τον κτηνοτρόφο. Δεν εφαρμόζεται λοιπόν η νομοθεσία και έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσκύψει πάνω στο πρόβλημα και να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα πριν το τέλος του 2016, το οποίο θα μας δείχνει πώς ακριβώς θα προχωρήσει και θα ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Δεν πρέπει να ε, ακούμε μόνο τους ε, και να ακούμε τις υποσχέσεις τους. Τα ζώα υποφέρουν εδώ και πάρα πολλά ε, χρόνια και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι πόσο επώδυνη είναι αυτή η πρακτική. Είναι καιρός λοιπόν να γίνει κάτι γι' αυτό και όπως ε, είπατε υπάρχει νομοθεσία αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία κρέατος το έχει συνειδητοποιήσει και θα συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, διότι το θέμα αυτό για την τακτική κοπή της ουράς των χείρων έχει συζητηθεί τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν. Είχαμε και την μελέτη της ε, Επιτροπής. Έχουμε στείλει επίσης και μια επιστολή στον Επίτροπο Αντριου Κάιτης για την πιθανότητα κινήσεις διαδικασίας επί παραβάση. Επίσης έχουμε ζητήσει και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να βάλει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, διότι συμμεριζόμαστε και εμείς τις απόψεις σας. Θέλουμε να δοθεί ένα τέλος αυτήν την ε, φρικτή πρακτική. Και συμμερίζομαι επίσης την άποψή σα ότι θέλουμε να δούμε και ένα χρονοδιάγραμμα δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει τις βέλτιστες πρακτικές όπου εντοπίστηκαν σε χώρες όπως η Φιλανδία για παράδειγμα, αλλά ας μην αρκεστούμε σε αυτό, ας αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες, ας αναλάβει κομισιόν τις ευθύνες της και ας δώσει επιτέλους ένα τέλος Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και ίσως να κάνει και έναν απολογισμό, μία εκτίμηση της κατάστασης στα κρατημέλη. Ποια από αυτά συμμορφώνονται πλήρως με την νομοθεσία, ποια από αυτά διστάζουν, ποια από αυτά την παραβιάζουν κατάφορα. Θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό. Μετά, εμείς από την πλευρά μας θα μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και να κλείσουμε την αναφορά. Όχι όμως προτού εσείς μας παρέχετε τις πληροφορίες που έχουμε ζητήσει. Μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχω την εντολή του Σώματος των Επιτρόπων για να κάνω μια τέτοια δήλωση, όπως καταλαβαίνετε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να εργαστούμε. Πρόεδρος, καλώς. Ωραία. Τότε τελειώσαμε και με αυτές τις αναφορές και περνάμε στην επόμενη αναφορά που είναι επίση για τα ζώα. Πρόκειται για τους σκύλους στην Φιλανδία. Δεν είναι εδώ η αναφέρουσα. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκληρά δουλεύετε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, παρακαλώ, για την αναφορά 1071 της Λίντα Μάκη Σούλκαβα όσον αφορά την αναπαραγωγή μη υγιών χαρακτηριστικών σε ζώα. Ποιος θα πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Υπάρχει κάποια σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Okay, so... Καλώς. Υποθέτω ότι υπάρχει κάποιο μπέρδεμα στην Επιτροπή και κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο για την αναφορά αυτή. Σωστά. Τότε, οι συνάδελφοι, έχετε δει την αναφορά, την έχετε μελετήσει προσεκτικά φαντάζομαι. και έχετε και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου βέβαια είναι στους φακέλους σας, οπότε μπορείτε να το κοιτάξετε και αυτό. Ωραία, ποιος θέλει το λόγο. Γενναιόδωρα. Έδωσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκολουθεί αν θέλει να πάρει το λόγο ευχαρίστω, αλλά και συνάδελφοι, οποίο συνάδελφος θέλει να συμμετάσχει ευχαρίστω επίσης. Κανεί δεν έχει να πει τίποτα από ό,τι βλέπω. Α, ο Πίτερ. Σε γενικέ γραμμέ να πω ότι η εκτροφή ζώων τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να αναπαράγει επιθυμητά χαρακτηριστικά σε αυτά τα ζώα. Αυτό μπορεί να είναι ε, κάτι το θετικό, κάτι το αρνητικό. Υπάρχουν και κάποιοι εκτροφείς της πλάκας, θα έλεγα, οι οποίοι δεν παίρνουν τα σοβαρά και ε, τη, δουλειά τους και δεν συμμορφώνονται με τα ε, πρότυπα της σωστής συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε για σκύλους και ορισμένες ράτσες που πρέπει να έχουν κάποια επιθυμητά, σύμφωνα με κάποιους που κάποτε το αποφάσισαν, χαρακτηριστικά. Ε, θα ήθελα λοιπόν εδώ να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σχετική μελέτη, τι γίνεται, που να μπορούμε να συνδυάσουμε με αυτήν την αναφορά. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω πως το θέμα είναι κοινωνικοπολιτικό και πρέπει να δούμε πού θα μπει το όριο ανάμεσα στην εκτροφή ζώων και το φασανισμό ζώων. Όταν ε, ο άνθρωπος, ξέρετε, δημιουργεί διάφορα ε, τέτοια ε, χαρακτηριστικά στα ζώα, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτό είναι σωστό και ηθικό και πρέπον. Ο άνθρωπος σίγουρα δεν θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για τα οποία είναι ικανός. Και σίγουρα Κανείς δεν ρωτάει το ζώο εάν αισθάνεται καλά με αυτά τα χαρακτηριστικά που ε, του έδωσαν. Και μια που μιλάμε για σκύλους, σίγουρα θα έχετε δει όλοι σας σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ε, είδατε γιατί έχει κάνει ο άνθρωπος από ένα λύκο. Πόσες διαφορετικές μορφές σκύλου έχει φτιάξει. Ωστόσο, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς να ξέρουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Γι' αυτό ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ε, μελέτες για να δούμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Και επίσης, επαναλαμβάνω, να κάνουμε και το διαχωρισμό ανάμεσα στην εκτροφή, ε, τη σοβαρή εκτροφή ζώων και τους βασανιστές αυτών. Πάντως σίγουρα το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο και πρέπει να συζητηθεί γιατί δεν αφορά μόνο τους σκύλους. Ευχαριστώ. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα ενημερωμένη για το θέμα αυτό, διότι αν διαβάσετε το συνοδευτικό έγγραφο έχουν αποφασίσει να εκπονήσουν μία μελέτη για την ευθορία σκυλιών και γατιών. Και στόχος είναι η αξιολόγηση του αν ε, αυτές οι ανησυχίες αποτελούν μια γενικότερη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Πίτερ να σε ενημερώσω ότι δεν θα γίνει μελέτη, έγινε μελέτη και δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2015. Γι' αυτό λοιπόν εσύ δεν είσαι καλά διαβασμένος. Και δεδομένη της μελέτης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα εξετάσει, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που διαβάζω, εάν χρειάζεται περαιτέρω δράση που ε, θα σχετιστεί με τις αρχές της επικουρικότητας και της αλλαλογικότητας. Εγώ προτείνω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και καλώ την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες να ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και θα ήθελα εδώ να σας παρακαλέσω ευγενικά να επανέλθετε πριν το τέλος του 2016 στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά και να την κλείσουμε. Συμφωνούμε? Μα τι έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Και τώρα σε αυτό το σημείο νομίζω πως ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Αλλά μισό λεπτό, μισό λεπτό κυρία Στανόκα. Μια και νωρίτερα εξετάσαμε το σημείο 16, την αναφορά δηλαδή 2453 από την Νάνση Σχάουτεν για την απομάκρυνση των παιδιών της από τις Σουηδικές ε, Αρχές Παιδικής Μέριμνας. Ε, να πω ότι η αναφερόμενη δεν ήταν παρούσα, ήρθε όμως τώρα μαζί με τα δύο της παιδιά και θα σας ενημερώσω, κυρία Σχάουτεν, για το τι συνέβη. Η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την αναφορά. Δεν γίνεται λοιπόν να ανοίξει πάλι. Έχει κλείσει η αναφορά και αν έχετε κάποια αλλά παράπονα πρέπει να υποβάλλεται νέα αναφορά. Εδώ είμαστε θεσμικό όργανο και όχι ε, κάποια ανεπίσημη παρέα σε μία λέσκη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Πρέπει να ακολουθηθούν οι επίσημες διαδικασίες. Ωστόσο θα σας δώσω το λόγο για να συνοψίσετε το τι έγινε μια που καθυστερήσατε να έρθετε την ώρα που εξεταζόταν η αναφορά σας και να κάνετε κάποια δήλωση σχετικά με αυτή. Έχει κλείσει η αναφορά, γι' αυτό λοιπόν δεν θα την ξανανοίξουμε. Σας ενημερώνω. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι. Έφτασα. Το κατάλαβα αυτό που είπατε, ότι είναι έχει κλείσει πια, αλλά θα ήθελα να σας πω την απόψή μου για το τι έγινε το καλοκαίρι του 2013 από τις ε, αρχές της Σουηδίας. Ξεκίνησε πολύ ωραία το καλοκαίρι μας, ε, πήγαμε στο ζωολογικό κήπο, σε άλλα μέρη και μετά πάρα πολλές κατηγορίες ε, ψευδείς από διαδόσεις των γειτόνων ε, ή των αρχών έκαναν τη ζωή μας κόλαση. Είπαν ότι δεν είχαμε νερό, ηλεκτρισμό, ούτε αρκετό φαγητό στο σπίτι. Και μετά τον ε, Ιούλιο οι αρχές μπήκαν στο σπίτι μας. Εμείς τους δείξαμε ότι ούτε είχαμε κλειδώσει τα παιδιά μας, ότι είχαν να παίξουν παιδική χαρά εκεί στην αυλή και ότι είχαμε και ηλεκτρισμό και τρόφιμα και απ' όλα και νερό. Τους δείξαμε και τους λογαριασμούς που πληρώναμε, την τουαλέτα μας, ε, τα δύο μπάνια. Αλλά αυτό δεν έκαναν καμία διαφορά σε αυτούς. Οι κοινωνικοί λειτουργοί πήραν και τα πέντε παιδιά, ακόμα και την μεγάλη μου κόρη, 19 ετών, χωρίς να εξηγήσουν, να μας μεταφράσουν κάτι. Απλώς εφάρμοσαν το σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους. Κατά από άνθρωπες συνθήκες λοιπόν τα παιδιά χωρίστηκαν και βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της Σουηδίας. Και εγώ δεν είχα δικαίωμα να τα επισκεφθώ για τρεις μήνες αρχικά και μετά για άλλους οχτώ. Έπρεπε να περιμένω. Δεν έπρεπε να είχε γίνει ότι έγινε. Εμείς δεν είμαστε Σουηδοί πολίτες ούτε τότε ούτε τώρα. Δεν βλέπω γιατί αναμίχθηκαν οι Σουηδικές αρχές. Σε ένα σωστό σουηδικό σύστημα και με τις αποδείξεις που είχα, είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να πάρω πίσω τα παιδιά μου, αλλά τελικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Σουηδία. Οι δικηγόροι, τα νοσοκομεία, οι δημοσιογράφοι, οι δικαστές, όλοι αυτοί συνεργάζονται για να κυκλοφορεί το χρήμα. Μετά την απόφαση, τρία από τα μεγαλύτερα παιδιά μου μου επιστράφησαν. Τα δύο όμως πιο μικρά παρέμειναν στη Σουηδία σε ανάδοχους ε, διεφθαρμένους γονείς. Δύο στη Σουηδία, δύο ε, στη χώρα μου. Πού ξέρω τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Δεν έχουν μπορέσει καν να κρατήσουν τη δικιά τους την ταυτότητα. Τα χειραγώγησαν για να γίνουν, τους είπανε, καλοί Σουηδοί πολίτες και δεν τους επιτρέπουν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Οι ανάδοχοι γονείς μόνο για τα χρήματα ενδιαφέρονται. Πήραν πολλά χρήματα επειδή ασχολούνται με τα παιδιά μου. Στο μεταξύ τα παιδιά μου όμως εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους και καταχρήσεις και έχουν καταστραφεί συναισθηματικά. Ένα ολόκληρο χρόνο. Η κατάχρηση αυτή πρέπει να σταματήσει στη Σουηδία. Τα παιδιά μου έχουν κατασταθεί συναισθηματικά. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ελπίζω ότι όλος αυτός ο φόβος που περάσαμε, όλο αυτό το άγχος, η αγωνία, να μην τα περάσαμε για τίποτα. Να πιάσουν τόπο προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Και ευχαριστώ όσες υπηρεσίες με βοήθησαν ώστε να καταφέρω τελικά να πάρω πίσω τα παιδιά μου, αλλά όπως σας είπα συναισθηματικά καταστραμμένα. Πρέπει να σηκώσουμε όλοι το ανάστημά μας για μια δικαιοσύνη που λειτουργεί. Να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα και προστατευμένα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που είπατε. Ε, χάρηκα που καταφέρατε να φτάσετε στις Βρυξέλλες και ελπίζω ότι εσείς και τα παιδιά σας θα περάσετε καλά την ημέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι πάντα καλό να συναντάμε αυτοπροσώπως τους αναφέροντες, γιατί έτσι ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από έναν αριθμό αναφοράς. Σας ευχόμαστε κάθε καλό από την Επιτροπή μας, ένα happy end και να περάσετε ωραία την ημέρα εδώ. Σας ευχαριστούμε. Ωραία, τώρα σε εσά συνάδελφοι, ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί σήμερα το πρωί στη δουλειά μας. Μπορείτε να έχετε περισσότερο μεσημεριανό διάλειμμα. 3 η ώρα ακριβώς εδώ με τον Επίτροπο Τίμερμανς.